Dear colleagues. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας. Πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσια διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες αυτή τη στιγμή και ως συνήθω. Οι φάκελοι της συνεδρίασης και τα κείμενα είναι διαθέσιμα μέσα της εφαρμογής e-meeting και επίσης θα μεταδοθεί από το διαδίκτυο. Στο σημείο 3 να ενημερώσω την Επιτροπή για το αποτέλεσμα του τρομερού διαλόγου για τη ιατροτεχνολογικά και τις διαγνωστικές ε, in vitro συσκευές. Ο έβδομος γύρος έλαβε χώρα στις 16 Μαρτίου 2016. Ήταν ο δεύτερος τρίλογος επί, τριμερής διάλογος επί Ολλανδικής Πρεδίας, όπου αποφασίστηκαν κάποια σημαντικά πολιτικά σημεία. Η τελευταία συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου που υιοθετήθηκε από το κορεπέ στις 9 Μαρτίου για τα θέματα της επανεπεξεργασίας, του ελέγχου για τα ιατροτεχνολογικά υψηλού κινδύνου, τις ε, ουσίες CMR, την ε, αξιοπιστία και το αίσθημα ειδοποίηση για τα φάρμακα εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο μαζί με το άρθρο 26. Το θέμα του ελέγχου για τι in vitro συσκευέ ακόμη δεν έχει επιληθεί. Το Ευρωκοινοβούλιο υποέβαλε τη θέση του για συγκεκριμένε κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ ε, πράξει και τι διατάξει του, όπω επίση και τι συστηματικέ εκθέσει ασφάλεια της κατηγορίας 6, 19 και 21 με την μόνιμη εμπειρογνωμοσύνη από τις εθνικές αρχές και των υπευθύνων φορέων in-house. Ε, ο επόμενο γύρος θα γίνει στι 7 Απριλίου. Και τέλο το θέμα τη γενετική συμβουλευτική για τι in συσκευέ συζητήθηκε ξανά στο Συμβούλιο, όπου επαναλήφθηκαν οι περιορισμοί τη θέση του Συμβουλίου για το σημείο αυτό. Το επόμενο σημείο, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διασυνοριακές συνέπειες των περιβαλλοντικών μελετών αντικτύπου. Όπως θα θυμάστε, είχαμε συζητήσει το σημείο αυτό μετά από αίτηση του Χέλμουτ Βόλφλεμ ο οποίος ε, ε, υπέβαλε την αναφορά 1555 στα γερμανικά και τσεχικά σύνορα και βάσει της απόφασης της 1ης Δεκεμβρίου 2015. Αποφασίσαμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δώσω λόγο στην, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, αρχική εισήγησή της στον κύριο Κρέμλης από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Παρακαλώ, έχετε το λόγο για την ομιλία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σε αδερές γραμμές τη διαδικασία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Στα αριστερά της διαφάνειας έχετε την οδηγία για τις ε, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ε, δεξιά την σύμβαση ΕΣΠΟ για τα διασυνοριακά σχέδια που έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το άρθρο 7 καλύπτει τα διασυνοριακά αποτελέσματα και την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση που κάποια σχέδια έχουν τέτοιες διασυνοριακές ε, συνέπειες. Έχουμε το παράρτημα 1 με υποχρεωτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεδομένων ε, των σχεδίων που υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε και το παράρτημα 2 στην οδηγία, όπου είναι προαιρετική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια που δεν είναι τόσο σημαντικά από άποψη περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και αντικτύπου. Αλλά συνήθως χρειάζεται ένα είδους ε, διεξοδικός έλεγχος. Πάμε στα δεξιά τώρα της διαφάνειας. Ε, η σύμβαση ΕΣΠΟ τέθηκε σε ισχύ το 1997. Είμαστε συμβαλόμενα μέρη στη σύμβαση ΕΣΠΟ. Αποκινούμε τα κράτη-μέλη. Το παράρτημα 1 παρουσιάζει ένα κατάλογο δραστηριοτήτων που υπόκειται στην υποχρέωση μελέτης επιπτώσεων δυνάμει της σύμβασης ΕΣΠΟ. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ε, διακυβερνητικό χαρακτήρα και διεθνούς δικαίου. Η υφιστάμενη οδηγία για τις ε, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων τροποποιήθηκε από τη νέα οδηγία 2014-52 που αντικαθιστά την προηγούμενη και που αναμένεται να ακυρωθεί από τα κράτη-μέλη του χρόνου και άρα να τεθεί σε εφαρμογή του χρόνου, ε, γιατί ήδη είναι ενισχύ. Η οδηγία 92 του 2011 έχει τροποποιηθεί και προβλέπεται η σύσταση ενός ε, κοινού φορέα για να εξασφαλίσει τη διαδικασία συντονισμού σε περίπτωση εκτίμησης επιπτώσεων ε, για σχέδια διασυνοριακού χαρακτήρα, με διασυνοριακές συνέπειες, ε, κάτι που προϋποθέτει διαβουλεύσεις που πρέπει να γίνουν σε πολλά κράτη-μέλη. Και φυσικά και ο αντίκτυπος ε, θα επηρεάζει τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Οπότε τα, τα ενδιαφέρομενα κράτη-μέλη μπορούν να συστήσουν ένα κοινό φορέα για το συντονισμό αυτή τη διαδικασία. Το σημαντικό είναι ότι η δυνάμη τη νέα οδηγία προβλέπεται η δυνατότητα εξορθολογισμού των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή προβλέπεται η δημιουργία μονοπευθυντικής θηρίδας, one stop shop, οπότε οι εκτιμήσεις αυτές και δυνάμει της οδηγίας για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και η εφαρμογή ε, τις πλαίσιο για το ή για τα οικοσυστήματα να υπόκεινται σε συντονισμό ή να περιλαμβάνονται σε μια κοινή διαδικασία εκτίμηση επιπτώσεων. Η σημασία της ε, διαδικασίας της οδηγίας για τις μελέτες επιπτώσεων καταρχήν εξασφαλίζει πολιτική και κοινωνική λογοδοσία και άρα καθιστά πιο αποδεκτή κοινωνικά τα σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη. Πρόκειται για ένα νομοθετικό μέσο που ε, προβλέπει διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, παροχή πληροφοριών και άρα ε, ενισχύει την κοινωνική αποδοχή σημαντικών project, σημαντικών σχεδίων και επίσης ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης που προβλέπουν τέτοιου είδου ε, δημόσιε διαβούλευση συμμετοχής ε, και ενημέρωσης. Μάλιστα, η οδηγία αυτή έχει τη ερμηνεία και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε σημαντική νομολογία από αυτού. Και επιπλέον η διαδικασία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κάτι που με βάση και το Διεθνές Δικαστήριο έχει αναγνωριστεί ως αρχή εθιμικού δημοσίου διεθνούς δικαίου. Τώρα, διασυνοριακά σχέδια που απαιτούν τέτοια, τέτοια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουμε την περίπτωση όπου έχουμε ένα μέρος προέλευσης, ένα συμβαλόμενο μέρος προέλευσης, δηλαδή τη χώρα στην οποία λαμβάνει η χώρα το σχέδιο, το project, την δραστηριότητα και είναι οι περισσότερα θυγόμενα μέρη, δηλαδή ένα, οι περισσότερα κράτη-μέλη όπου βιώνονται οι συνέπειες των σχεδίων, των project, των δραστηριοτήτων του συμβαλόμενου μέρους προέλευσης. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για project που έχουν διασυνοριακά αποτελέσματα και αντικτύπωση περισσότερο από ένα μέρος, συμβαλόμενο μέρος προέλευσης και περισσότερο από μία θυγόμενη χώρα μέλος. Πρόκειται για σχέδια που αποκαλούμε διασυνοριακά σχέδια μεγάλης κλίμακος ή μεγάλης εμβέλειας. Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση ΕΣΠΟ που ε, ισχύει για τα κράτη-μέλη, όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλα όσα την έχουν κυρώσει. Μπορεί να ε, υπάρχουν κάποια σχέδια που αναπτύσσονται το, μεταξύ χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΣΠΟ, αλλά ε, μέλη της σύμβασης αυτής, μέρη της σύμβασης αυτής είναι θυγόμενα μέρη Είχαμε μια περίπτωση το Nord Stream 1 που χώρα προέλευσης ή ή μέρο πρόελευσε η μερο προελευση ηταν η ρωσια που δεν έχει προσυπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΟ αλλά de facto και τι ανάγκε του σχεδίου Nord Stream έχει υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, υλοποιούν, δεν πρέπει να καταρτίζουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είναι ούτε συμβαλωμένο μέρος προέλευσης ή ούτε θυγόμενο μέρος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μόνο τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι συμβαλωμένα μέρη προέλευσης ή θυγόμενα μέρη. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όπως εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι ούτε μέρος προέλευση ούτε θυγόμενο μέρος. Και αυτό με βάση τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Φυσικά, εμείς ως θεματοφύλακες της συνθήκης ε, ε, έχουμε το καθήκον να ελέγξουμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και φυσικά στο ευρωπαϊκό, στο κοινοτικό κεκτημένο εμπίπτουν και η οδηγία για τις ε, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η σύμβαση ΕΣΠΟ. ΕΣΠΟ. Τώρα, κάποιες ιδέες και πιθανές λύσεις. Συμμόρφωση ε, με την εφαρμοστή νομοθεσία και εφαρμογή της που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από όλα τα συμβαλόμενα μέρη που συμμετέχουν σε διασυνοριακά project σχέδια. Αυτή είναι η ευθύνη τους. Τα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να μεριμνήσουν ε, για την εφαρμογή και συμμόρφωση με το κοινό κεκτημένο. Καλή και επικοδομητική ε, επικοινωνία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών επίσης είναι πολύ σημαντική. Συντονισμός και συνεργασία απαραίτητα στοιχεία. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια κατευθυντήρια έγγραφα και οι διμερείς συμφωνίες ε, υπό την Σύμβαση ΕΣΠΟ για να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα βλέπετε στα κατευθυντήρια αυτά έγγραφα, έχουμε ένα έγγραφο για τη διαδικασία περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλης κλίμακος διασυνοριακά σχέδια. Το βλέπετε αριστερά της οθόνης. Υπάρχει αυτό το έγγραφο στο, συγκεκριμένο link και επίσης ε, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για υποδομές ενέργειας και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Για αυτά τα δύο σημεία έχουμε ήδη τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά εισαγωγικά και είμαστε στη διάθεσή σας κύριε Πρόεδρε για να λύσουμε τις απορίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε τώρα την συζήτησή μας. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπατε στην αρχή κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση σχετίζεται με μία αναφορά. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μία περίπτωση με διασυνοριακές επιπτώσεις, τότε όλα είναι εντάξει. Αλλά ε, ποιος αποφασίζει αν υπάρχουν εδώ διασυνοριακές συνέπειες. Ε, εδώ έχει συμβεί το εξής. Οι Τσέχοι έχουν ε, χτίσει στη Γερμανία αιωλικό πάρκο και είπαν ότι στα σύνορα εντός της Τσεχίας ε, και είπαν ότι αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη Γερμανία. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις τότε δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να ενημερώσει για κάτι. Ποιος ε, διαπιστώνει εάν υπάρχουν ε, διασυνοριακές επιπτώσεις. Ε. Να σας πω τη δική μου γνώμη. Δεν μπορεί ο ανάδοχος να λέει από μόνος του ότι εγώ διαπιστώνω ότι το δικό μου έργο δεν έχει επιπτώσεις στον γειτονά μου, στη γειτονική μου χώρα. Θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνω τον γείτονά μου σε τέτοιες περιπτώσεις ε, και ακριβώς γι' αυτό ε, έχει υποβληθεί η αναφορά αυτή. Εάν λοιπόν ε, διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, υπάρχει μια πολύ ωραία διαδικασία, αλλά το πρόβλημα εδώ είναι στο στάδιο πριν από αυτό. Διότι από την αναφορά προκύπτει ότι η Τσεχία είπε ότι «Α, συγγνώμη, δεν σα ενοχλεί καθόλου ε, το έργο μου και έχω εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων». Το θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ποιος αποφασίζει αν υπάρχουν διασυνορικέ επιπτώσεις. Η κυρία Πύρικ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία έμεση ερώτηση μάλλον. Στην Ευρώπη έχουμε επίσης και την οδηγία περιπτυνών. Ε, τα κράτη-μέλη εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Στις κάτω χώρες σίγουρα εργαζόμαστε πάνω στο θέμα. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Χόχφεν που βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα. Εκεί υπάρχει ένα είδος τύρφης και αναρωτιόμαστε εάν θα πρέπει να προστατεύσουμε τις περιοχές αυτές. Αυτό αφορά και τις εκμεταλλεύσεις. Κατά την εξαγωγή λοιπόν αυτού του προϊόντος θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Διότι σε κάποιες χώρες επιτρέπονται κάποια πράγματα, σε άλλες χώρες όχι. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει διαδικασία για να αποφεύγουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κονέτσινα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η οδηγία σε γενικές γραμμές δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και πρέπει να πω ότι και για το κοινό, και για το κοινό της χώρας μας ε, Okay. Thank you very much. Já bych chtěla jenom upozornit na to, že implementaci této směrnice došlo και πάλι να πω ότι η υλοποίηση της οδηγίας ε, δεν γίνεται σωστά, γιατί θα έπρεπε να ισχύει για διαφορετικές απειλές όμως εμείς ως νομοθέτες από την Τσεχία μπορέσαμε να επιλύσουμε την κατάσταση στη δική μας χώρα και να μεταφέρουμε την οδηγία σωστά. Όμως πιστεύω ότι είναι πολύ, περιοριστική, πολύ περιοριστικός ο κατονισμός που έχουμε. Είναι από τους πιο περιοριστικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δυσκολεύει όσους ε, αναπτύσσουν τα προγράμματα, όσους τα εκπονούν και πραγματικά έχει τους ευρύτατους, ευρύτατες συνέπειες η νομοθεσία που προβλέπουμε. Οι επενδυτέ μα λοιπόν μα λένε ότι καμιά φορά θέλουν να φύγουν από την Τσεχία να πάνε στη Γερμανία να επενδύσουν, διότι βάσει τη γερμανική νομοθεσία μπορούν να πάρουν τι άδειε που θέλουν και τι εξουσιοδοτήσει μέσα σε ένα τρίμηνο. Ενώ στη δική μα τη χώρα χρειάζονται τρία, πέντε ή και καμιά φορά δέκα χρόνια για να πάρει κανεί άδεια. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, μια και είναι εδώ εκπρόσωπο τη Επιτροπή, και να πω. Το εξή, ήθελα να ρωτήσω, δεν θα άξιζε να υπάρξει εναρμόνιση αυτών των κανόνων σε όλη την Ευρώπη, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιβάλλει διαφορετικού όρου και προποθέσει στα διάφορα κράτη-μέλη και να μην αποφασίζει για το τι θα ισχύει στην χώρια νομοθεσία. Πιστεύω ότι σήμερα, ε, έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσει, δεν έχουμε ισοκανονισμού κανόνε παιχνιδιών, δεν υπάρχει ισοτιμία και δίκαιο ανταγωνισμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ αυστηρότερη με τι ε, μικρέ χώρε αλλά όχι με τι μεγαλύτερε. Καταλαβαίνουμε το νόημα και το σκοπό αυτή τη οδηγία, όμω η υλοποίηση και η μεταφορά τη στι επιμέρου χώρε μέλη είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όλο αυτό μα οδηγεί σε καταστάσει όπω αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα η αναφορά, η αναφορά που τώρα εξετάζουμε, αυτού του Γερμανού πολίτη που ε, παραπονείται για τα τσεχικά προγράμματα. Όμως παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα κρατημέλη, ακριβώς γιατί δεν έχουμε καταφέρει να συντονίσουμε τους κανόνες μας. Δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα από τις ε, περιβαλλοντικές μελέτες αντικτύπου. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εάν ε, μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Οδηγία για να γίνουν επιτέλου ισότιμοι κανόνε του παιχνιδιού για όλα τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Να τους ζητήσουμε να μας απαντήσουν. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά. Και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ποιος καθορίζει κατά πόσο ένα σχέδιο έχει διασυνοριακές συνέπειες. Υπάρχει μια διαδικασία κατά την οποία ο ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει μια περιβαλλοντική έκθεση με μια τεχνική σύνοψη και με εκτίμηση όλων των πιθανών επιπτώσεων του project. Και πολύ συχνά η περιβαλλοντική έκθεση έρχεται μετά από το αίτημα που κάνει ο ανάδοχος προς τις αρμόδιες αρχές να καθορίζουν το πεδίο εφαρμογή και το επίπεδο πληροφοριών που οφείλει να συγκεντρώσει για να συμπεριλάβει στην περιβαλλοντική του έκθεση. Οπότε, το εργαλείο για να αποδείξουμε το διασυνοριακό χαρακτήρα και το διασυνοριακό αντίκτυπο είναι η περιβαλλοντική έκθεση. Πολύ συχνά όμως έχει γίνει πρώτα μια ανάλυση του πεδίου εφαρμογή. Ιδιαίτερα για περίπλοκα σχέδια, για να είναι καλυμμένος ο ανάδοχος, θέτει ήδη ε, την ερώτηση στις αρμόδιες αρχές για το πεδίο εφαρμογής. Και συνήθως ε, οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν αν ε, υπάρχουν διασυνοριακά αποτελέσματα λόγω της ιδιαιτερότητας του σχεδίου. Αν έχουμε για παράδειγμα ένα σχέδιο που περνά τα σύνορα δύο χωρών, αν πρόκειται για έναν αγωγό, για παράδειγμα, ή βρίσκεται πολύ, συχνά, πολύ κοντά στα σύνορα άλλου κράτους μέλους και άρα κατά πάσα πιθανότητα θα έχει συνέπειες στο άλλο. Τώρα το επίπεδο πληροφορίας ε, και λεπτομέρειες της πληροφορίας βρίσκεται στο, στην περιβαλλοντική έκθεση που καθορίζει τα, τα διασυνοριακά αποτελέσματα και συνήθως υπόκειται στη γνωμοδότηση των περιβαλλοντικών αρχών και σε δημόσια διαβούλευση που μπορεί να είναι διαφορετικές από τις ε, αρμόδιες αρχές και καθορίζει κάποιες άλλες, κάποιες άλλες πτυχές που θα πρέπει να εκτιμηθούν. Αυτή είναι η διαδικασία και αν το κράτος μέλος κρίνει στη διαδικασία αυτή υπάρχουν διασυνοριακές συνέπειες, οφείλουν να το κοινοποιήσουν στέλνοντας κατάλληλες πληροφορίες στις θυγόμενες χώρες, που συχνά είναι οι γείτονες χώρες, οι όμορες χώρες. Υπάρχει όμως και άλλη πιθανότητα. Αν η θυγόμενη χώρα κρίνει ότι το σχέδιο που θα διεκπαιρεωθεί σε γειτονικό κράτος μέλος, για το οποίο η διαδικασία δεν προβλέπει διασυνοριακά αποτελέσματα, η θυγόμενη χώρα μπορεί παρόλα αυτά να πει ότι κρίνει ότι θα υπάρξουν τέτοια διασυνοριακά αποτελέσματα και άρα να απαιτήσει κοινοποίηση. Οπότε θα λάβει χώρα αυτή η διαδικασία κοινοποίησης με πληροφορίες και τις δημόσιας γνωμάτευσης ε, ή μάλλον των δημόσιων διαβουλεύσεων και στη θυγόμενη χώρα. Και μάλιστα η νέα οδηγία προβλέπει ότι οι διαβουλεύσεις για τα διασυνοριακά αποτελέσματα μεταξύ της χώρας προέλευσης και της θυγόμενης χώρας μπορούν να γίνουν από το κατάλληλο κοινό φορέα που θα συσταθεί ad hoc. Οπότε υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να ληφθούν υπόψη τα διασυνοριακά αποτελέσματα ενός σχεδίου. Ακόμη και αν δεν εντοπιστούν από τη χώρα προέλευση, μπορεί να εντοπιστούν από τη θυγόμενη χώρα. Οπότε ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 7 της νέας οδηγίας για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση της Ευρωβουλευτής από την Τσεχία, η οδηγία δεν χρειάζεται να ενσωματωθεί στην εσωτερική νομιτάξη με μαξιμαλιστικό τρόπο. Εμείς θέλουμε απλώς να μεταφέρονται σωστά στην εθνική νομοθεσία διατάξει της οδηγίας. Και αν ένα κράτος μέλος θέλει στην νομοθεσία εφαρμογή να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα, έχει τη διακριτική ευχαίρεια να το κάνει. Δεν είναι κάτι όμως που εμείς το ζητούμε από τα κράτη-μέλη. Να εθετήσουμε μια διασταλτική εφαρμογή δηλαδή της οδηγίας. Και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, εμείς ελέγχουμε τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της οδηγίας. Αυτές είναι που θα πρέπει να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία. Είχαμε κάποια προβλήματα με τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό τσεχικό δίκαιο, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το θέμα τώρα. Υπάρχει και αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση που προβλέπετε, γιατί η διαδικασία EA για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με χρηματοδότηση σε οποιοδήποτε σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η νέα οδηγία έχει ήδη εγκριθεί. Πρόκειται για την οδηγία του 2014 που αντικαθιστά την προηγούμενη του 2011 και πρόκειται για μια οδηγία που δεν είναι ακόμη ε, εφαρμοστέα. Τα κράτη-μέλη οφείλουν μέχρι το Μάιο του 2017 να, τα, να τη μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία Οπότε υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθεί νωρίτερα στην Εθνική Νομοθεσία πριν την καταληκτική προθεσμία του Μαΐου του 2017 και έτσι να διορθωθούν κάποιες αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο παρελθόν ή κάποιες διαδικασίες που θεωρώνταν ιδιαίτερα γραφειοκρατικές και επαχθείς για τους αναδόχους, για την προώθηση των projects τους. Πάντω η νέα οδηγία προβλέπει εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Οπότε, όπου ισχύουν πολλέ οδηγίε, το κράτος μέλο έχει επιλογή όταν μεταφέρει ε, το, τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο να προβλέψει είτε ε, κοινή είτε συντονισμένη μελέτη. Οπότε χρειάζεται μια δημόσια διαβούλευση και μια περιβαλλοντική έκθεση και αυτό έχει πολλά πλονεκτήματα για την περαιτέρω έγκριση των διαφόρων σχεδίων. Και τέλος, απαντώντας στην ε, Ευρωβουλευτή από, τη Δανία, από την Ολλανδία, συγγνώμη, θα ήθελα να πω ότι είναι αλήθεια ότι σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα οικοσυστήματα και τα πτηνά, Όντως αυτές ε, οι δύο οδηγίες υπόκειται τώρα στη διαδικασία του refit. Και περιμένουμε την έκβαση πριν το καλοκαίρι ε, του 2016 ε, για, τον έλεγχό τους. Επίσης για τις περιοχές του Natura 2000 φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε τις παραμεθόριες περιοχές και αν κάποια διασυνοριακά σχέδια επηρεάσουν, επηρεάζουν ζώνες του Natura 2000 θα πρέπει να ε, υπαχθούν και στις οδηγίες για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στα άρθρα 16 και 4 τις οδηγίες ε, για τα οικοσυστήματα και τα πτηνά. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί όλα αυτά να υπάγονται σε μία ενιαία εκτίμηση επιπτώσεων που να Εκτιμά ταυτόχρονα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις ε, στη φύση. Σας ευχαριστούμε για τις ε, απαντήσεις σας. Και τώρα και πάλι ο κύριος Γιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, δύο περιπτώσεις εδώ πέρα στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ. Νομίζω ότι οι υποχρεώσεις ε, περί ε, δεν ε, είχαν πληρωθεί στην περίπτωση αυτή. Εάν κάποιος θέλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του θα πρέπει να γνωρίζει τι να κάνει. Εάν χτίσω πυρηνικό εργοστάσιο, αυτό διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά είναι πολύ εύκολο να τοποθετήσει κανείς ε, γρήγορα ανεμογεννήτριες. Ε, έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το ελικό πάρκο χωρίς να ενημερωθεί η γερμανική πλευρά, δεν ε, ήταν προστατευμένη περιοχή. Έτσι θεώρησαν οι Τσέχοι ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις για την γερμανική πλευρά. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε από ε, τις ε, περιπτώσεις αυτές. Ε, λέτε ότι με την κοινοποίηση μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος, εντάξει. Αν μου λέτε πάντως όμως ότι οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται από τη νέα οδηγία, τότε μπορώ να πάω σπίτι μου ήσυχος. Ευχαριστώ πολύ. Να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο στις περιοχές ε, Natura 2000. Μπορεί ένα έργο εκτός των περιοχών αυτών που να μην βρίσκεται καν κοντά στα σύνορα να έχει επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει κοινοποίηση, διότι μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά την ρήπανση του αέρα, ε, των υδάτων, των ποταμών. που ε, ε, εξορισμού είναι διασυνοριακή ρήπανση, η ρήπανση των ποταμών, εφόσον το ποτάμι περνάει από άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται σωστή μελέτη των επιπτώσεων και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η απόφαση που, ε, γίνεται με, που λαμβάνεται με την ολοκλήρωση της μελέτης επιπτώσεων Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη της το σύνολο του έργου και υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και για πρόγραμμα που θεωρήθηκε ότι δεν έχει διασυνοριακές επιπτώσεις ε, μπορεί στο στα δικαστήρια της χώρας ε, προέλευσης ε, να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο. συχνά όταν ε, ε, ρωτάτε κανείς ε, θέλετε να ενημερωθείτε, θέλετε να γίνει κοινοποίηση. η απάντηση μπορεί να είναι ναι, σας παρακαλώ να μας κοινοποιείτε ή όχι δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να σας καθησυχάσω ότι η οδηγία αυτή προβλέπει όλα τα μέτρα ώστε να αποφευθούν τέτοιες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Α, ζήτω συγγνώμη, κυρία Κάντεμπαχ. Δεν είχα ζητήσει αρχικά το λόγο, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο REFIT, σε συνδυασμό με την οδηγία Περιπτεινών, θα ήθελα να σας θυμίσω τη θέση του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό για μας να γίνεται σωστή η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. και πιστεύουμε ότι άνοιγμα της σα νομοθεσίας ε, θα οδηγήσει ακριβώς στο αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Εμείς θέλουμε διατήρηση της βιοπικιλότητας. Αυτή ακριβώς είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα το κλείσιμο της υπόθεσης αυτής ε, και κατόπιν θα σας ε, ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε αυτό να συμβεί σύντομα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα έχουμε μια κοινή συζήτηση για το σημείο 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης. Είναι δύο ενστάσεις βάσει του άρθρου 106 για την ε, είναι ανανέωση της έγκρισης για την ε, δραστική ουσία γλυφωσοφ... Εδώ λοιπόν ξέρετε ότι για να θεωρηθεί παραδεκτή η αντίρρηση πρέπει να συνυπογραφεί από 30 τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ και τώρα έχουμε και από κάθε πολιτική ομάδα να υποστηρικτή αυτή τη αντίρρηση. Γι' αυτό να ξεκινήσω ευθύ αμέσω, δίνοντα το λόγο στον Πάβελ Πότ εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στην κατάρτιση του ψηφίσματος. Το κείμενο στηρίζεται στη δική μου πρόταση, γι' αυτό και θα μιλήσω λίγο περισσότερο από τους άλλους ε, συντάκτες η, η διαδικασία της κοινοβουλευτικής αντίρρησης είναι η, το ίστατο μέτρο που έχουμε, η άσχατη λύση και μάλιστα δεν είμαι υποχρεωμένη να καταφύγουμε καν σε αυτήν γιατί όταν καταφεύγουμε σε αυτή τη διαδικασία σημαίνει ότι κάτι πήγε στραβά ή ότι η όλη διαδικασία επιτροπολογίας που χρησιμοποιείται για την έγκριση ή επανέγκριση κάποιων δραστικών ουσιών είναι ελαττωματική ή κάπου ε, είχε προβλήματα. Από το 2012 που είχαμε την αρχική πρόταση είχαμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε και αναζωπηρώθηκε η συζήτηση πριν από ένα μήνα. Το Μάρτιο συμμετείχαμε σε μια διεθνή διάσκεψη όπου συμμετείχαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Ασφάλειας των Τροφίμων και ο Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία από τον Καρκίνο. Ε, φαντάζομαι όσοι συνάδελφοι δεν έδωσαν το παρόν δεν ενδιαφέρονται για τα επιστημονικά πορίσματα. Πάντω, μετά την ακρόαση αυτή, στείλαμε επιστολή στον κύριο Δρουκάητη ζητώντα αναβολή τη ψηφοφορία στην, επίσημη, στην ε, μόνιμη επιτροπή. Κάτι που συνέβη. Γιατί μετά από διαβουλεύσει και με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν συγκέντρωνε την ενισχυμένη πλειοψηφία που χρειαζόταν και άρα ανέβαλε την ψηφοφορία. Μάλιστα τον Ιούνιο εκπνέει η άδεια για την γλυφοσάτη και το Μάιο του 2016 θα συνεδριάσει και πάλι η μόνιμη επιτροπή. Παρόλο που έγινε περιορισμένες ερμοδιότητες για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω να λάβει στα σοβαρά ε, την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναθεωρήσει την πρότασή τη Εγώ ως γιατρός δεν δέχομαι την έγκριση μιας δραστικής ουσίας σε περίπτωση που οι επιπτώσεις δεν έχουν δεόντως αναλυθεί. Ιδιαίτερα αν μια τέτοια δραστική ουσία μπορεί να επηρεάσει το ενδοκρινολογικό σύστημα. Μάλιστα η γλυφοσάτη είναι μία από το κοκτέιλ δραστικών ουσιών στο οποίο εκτιθέμεθα. Ε, έχει κριθεί ως ε, δυνάμει καρκινογόνο από τον ε, αρμόδιο φορέα για την προστασία από τον καρκίνο του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Οπότε δεν θα πρέπει να ανανεώνεται η άδεια της δραστικής αυτής ουσίας άνεφόρων και μάλιστα αν οπωσδήποτε θα πρέπει να δοθεί άδεια θα πρέπει να είναι όσο πιο βραχία γίνεται και ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη τελευταίες επιστημονικές μελέτες προκειμένου να γίνει άμεση αναθεώρηση. Ερωτώ λοιπόν, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανταποκριθεί στη διαδικασία αντίρρησης που κίνησαν οι ευρωβουλευτέ. και δεύτερον, πώς ε, θα ε, συνεργαστείτε με την ΕΦΣΑ ώστε να δημοσιεύσετε τις ε, επιστημονικές μελέτες για το θέμα αυτό. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ανανέωση της άδειας για τη γλυφοσάτη για μία δεκαπενταετία, που είναι η μεγαλύτερη δυνατή περίοδο με βάση τη σχετική νομοθεσία. Λάβατε όμως απόψη την αρχή της προφύλαξης για την παράταση αυτή. Επίσης, ε, τι μέτρα λάβατε ώστε να οι να ελεγχιστοποιηθούν οι συνέπειες χρήσης της γλυφοσάτης. Πρόκειται να ελέγξετε ε, και να συνεχίσετε την παρακολούθηση των κατάλοιπων ε, γλυφοσάτης στη, στα τρόφιμα, όπως πρότεινε το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Καρκίνο. Η ΕΦΣΑ διατείνεται ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της είναι η μικροβιακή αντοχή. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνετε υπόψη το γεγονός ότι η γλυφοσάτη είναι και αντιβιωτικό. Μάλιστα καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αντιβιωτικό και συμβάλλει στη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιωτικά ενώ αποδεκατίζει την καλή χλωρίδα του εντέρου. Υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μελέτες που πιστοποιούν αυτά που σας λέω. Εξεπλάγει από το ότι στη συζήτηση που ακολούθησε στην Επιτροπή Γεωργίας αναφέρθηκαν πολλά το Μάρτιο. Εν κατακλεί θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα από αυτά Τα ανεξάρτητα εργαστήρια συνήθω διατείνονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τη γλυφοσάτη. Ενώ εργαστήρια που συνδέονται ή έχουν οικονομικά συμφέροντα με τον κλάδο παραγωγής τη ε, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κρίνουν ε, ανώδυνη τη γλυφοσάτη και ακίνδυνη. Η γλυφοσάτη βρίσκεται παντού είναι το πιο διαδεδομένο φυτοφάρμακο. Βρίσκεται στο έδαφος, στα τρόφιμα, στη γερμανική μπύρα που λατρεύω και που απολαμβάνω, που τουλάχιστον απολάβανα μέχρι τώρα. Και σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται η βιομηχανία, η γλυφοσάτη μεταβολίζεται πλήρως χωρίς ε, να αφήνει κατάλοιπα. Αυτός είναι ο ισχυρισμός της βιομηχανίας. Επίσης δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μελέτες ε, και συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερε μελέτε και συμφωνώ με το σχόλιο του κυρίου Δεκάστρο ότι μα λείπουν τέτοιε επιστημονικέ μελέτε εκτεταμένε. Ε, αναφέρθηκαν τρεις βασικές επιστημονικές μελέτες που πιστοποιούν τη σχετική κινδυνότητα της γλυφοσάτης, αλλά χρηματοδοτήθηκαν από την ε, βιομηχανία φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει ένας ανεξάρτητος φορέας να κάνει τις ε, σχετικές μελέτες και όχι μόνο για τη γλυφοσάτη, για οποιαδήποτε παρόμοια δραστική ουσία. Ο κύριος Ντέση είπε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε, σε επιστημονικά πορίσματα και όχι σε ιδεολογικά κριτήρια. Μα βεβαίω, αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς. Έγινε επιστημονική διάσκεψη, εγώ την οργάνωσα, μάλιστα απουσίασε από αυτήν ο γιατί αν είχε έρθει στην επιστημονική διάσκεψη θα είχε καταλάβει πολύ περισσότερα για την γλυφοσάτη. Αν εμεί ζητούμε επιστημονική γνώση και επιστημονικά πορίσματα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε όταν υποβάλλονται. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε από το King's College ε, ένα καθηγητή από τη Λιψία, ένα καθηγητή από τις Ηνωμένε Πολιτείες και όλοι μας ε, παρουσίασαν και την ε, βιοχημική δράση της γλυφοσάτης, ε, τον τρόπο που γίνεται η βιοσύνθεσή τους, αλλά και πώς επηρεάζει τη χλωρίδα και την πανίδα. Επίσης, μίλησε για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα χαμηλών δόσεων γλυφοσάτης, που ούτε καν αυτό δεν εξετάζει η ΕΦΣΑ. φαίνεται από μελέτες στις ΗΠΑ ότι η γλυφοσάτη συνδέεται και με την ανάπτυξη πολλών ασθενειών. Τέλος, η γλυφοσάτη είναι, είναι μια σημαντική ουσία για τη γεωργία. Και κάποιοι διατείνονται ότι το αλκοόλ και ο καπνός είναι ακόμη πιο τοξικά από τη γλυφοσάτη. Μα αυτά είναι ιδεολογικά σχόλια και δεν ξέρω σε τι επιστημονικές μελέτες ε, αναφέρεστε και σίγουρα η τοξικότητα του αλκοόλ μπορεί να είναι υψηλότερη από αυτή της γλυφωσάτης, αλλά το ίδιο ισχύει και για το αλάτι. Εδώ όμως μιλούμε για μια ουσία που επηρεάζουν το μεταβολισμό των κυτάρων ε, και μπορούν να διαταράξουν το ενδοκρινικό σύστημα. Επίσης ε, αναστέλει το CIP 450. Και ο παραλυσμός με την καφέινη και το αλκοόλ έχει κάποια βάση γιατί ε, δημιουργούν εθισμό και οι δύο ουσίες αυτές, αλλά πιστεύω ότι ειδικά για την γλυφοσάτη, αν, την αποσύρουμε από τη γεωργία, θα έχουμε πολύ πιο υγιεινά τρόφιμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κονέτσινα από την ΚΟΕ. Κυρίες και κύριοι, Ο κύριος Πότσο είναι ο κύριος που ξανανοίγει το θέμα. Ήδη μίλησε αρκετά για το θέμα, αλλά να σας κάνω μια σύντομη σύνοψη. Πριν από εννέα μήνες συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε την αντίρρησή μας όσον αφορά την επανέγκριση της γλυφοσάτης ως δραστική ουσία. Ε, απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τώρα Έχουμε την γνωμοδότηση, αλλά η γνωμοδότηση αυτή πιο πολλά ερωτήματα θίγει παρά δίνει απαντήσεις. Η διαδικασία φαίνεται πολύ περίεργη. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με το θέμα εδώ και πολύ καιρό, αλλά και το κοινό γενικά και μάλιστα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, έχουν εκπλαγεί πολύ δυσάρεστα σχετικά με το πώς χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση ε, ε, ε, φυτοφαρμάκων και ζυζανιοκτώνων. Και Όλο και περισσότερες μελέτες ε, δημοσιεύονται που δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι η ουσία αυτή για την ε, υγεία, για τα ε, υπόγεια ύδατα και πολλές διεθνείς οργανώσεις, η Greenpeace και άλλες, κάθε μέρα μας επισημαίνουν πόσο επικίνδυνη είναι η γλυφοσάτη για την ανθρώπινη υγεία. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κλείνει τα μάτια απέναντι σε όλες αυτές ε, τις αντιρρήσεις. Και είχα μια συνάντηση στο Στρασβούργο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ακόμα είμαι συγκλονισμένη όταν σκέφτομαι το πώς διεξήχθη αυτή η συνάντηση. Πρόκειται για καρκινογενή ουσία και παρόλα αυτά έγινε ανανέωση της άδειαση για την γλυφοσάτη για έξι μήνες. Οι συνάδελφοι είπαν ότι αυτό θα είναι το μακρύτερο χρονικό διάστημα ε, που θα μπορούσαν να δεχτούν, ε, εκτός εάν μπορούσε κανείς να διασκεδάσει τις ε, ανησυχίες τους. Αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά δυστυχώ η ΕΦΣΑ έχει χάσει την αξιοπιστία τη εδώ και πολύ καιρό. Και όχι μόνο λόγω της τελευταίας έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η ΕΦΣΑ ε, έχει εγκρίνει τη ζαχαρίνη που έχει απαγορευτεί στι Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά ε, επειδή είναι καρκίνογενή ουσία. Ε, υπάρχουν ουσίες που τις συζητάμε εδώ κάθε μήνα λόγω της συμφωνίας TTIP. Αρχικά λοιπόν μιλούσαμε για ε, επανέγκριση για ένα εξάμεινο, τώρα μιλάμε για 15 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για την υγεία των πολιτών της. Κυρίες και κύριοι, δεν πιστεύω ότι η δική μας ε, Επιτροπή θα πρέπει να δώσει την ευλογία της ε, στο θέμα αυτό. Είμαστε αρμόδιοι για την δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν, θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωση. Επιτροπής και της ΕΦΣΑ. Δεν ε, χρειαζόμαστε τέτοιες ε, ουσίες στην Ευρώπη, να μην ε, ευνοήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις εις βάρος των πολιτών μας. Η έγκριση χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια της ουσίας. Αν δεν ξέρουμε ποιον ε, να εμπιστευτούμε, ας εμπιστευτούμε τους εκλεγμένους ε, και ας εμπιστευτούμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να εξηγήσω στους συναδέλφους ότι ο κατάλογος των αγορητών Είναι πρώτα να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι των πολιτικών ομάδων που έχουν υπογράψει την αντίρρηση. Έπειτα οι άλλοι συνάδελφοι που δεν εκπροσωπούν πολιτικές ομάδες αλλά έχουν υπογράψει την αντίρρηση και μετά συνάδελφοι που δεν έχουν υπογράψει από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα. Για να εξηγήσω γιατί έχουμε αυτή τη διαφορετική ε, σειρά. Ο κύριος Στάις τώρα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η αντίρρηση αυτή όπως ξέρετε έχει, οφείλεται στην ε, τεράστια αύξηση χρήσης της γλυφοσάτης από το 1994, 160 φορές ε, περισσότερη χρήση σήμερα. Ξέρουμε ότι σε κάποια ζυζανιοκτώνα, σε κάποια φυτοφάρμακα παγκοσμίω χρησιμοποιείται κατά κόρον η ουσία αυτή και η γλυφοσάτη είναι Ε, μια ουσία που χρησιμοποιείται κατά τα τρία τέταρτα όλου αυτού του όγκου χρήση στα αγροτικά προϊόντα. Αλλά κάποιε φορέ και στα αυτοκίνητα και όλο και περισσότερο γλυφοσάτη έχουμε στο έδαφο, στο νερό, στα ε, τρόφιμα και αυτό ισχύει και, για την μπύρα που τόσο πολύ απολαμβάνει ο συνάδελφος, αλλά και στο μητρικό γάλα και στον αέρα που αναπνέουμε. Ε, ο άνθρωπος λοιπόν είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένος στην κλειφωσάτη σήμερα, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Βεβαίως, ο, οργανισμ, ο κανονισμός για τα φυτοφάρμακα του 2009 υποτίθεται ότι ε, επιλύει τα θέματα αυτά και μάλιστα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ε, και ένας νόμος του 2009 λέει ότι μπορούν ε, να εγκριθούν οι χρήσεις της γλυφοσάτης όταν δεν υπάρχει μεγάλη έκθεση των ανθρώπων σε αυτή ή όταν υπάρχει απαραίτητη προστασία της υγείας των φυτών ή άλλος διαφορετικός τρόπος για να την πετύχουμε αυτή δεν υπάρχει. Σε αυτό το νόμο του 2009 λέγεται ότι αναμένεται έγκριση της ε, ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Έχουμε βεβαίω πολλέ αντιρρήσει ω προ αυτό, αλλά ε, επίση προβλέπετε ότι η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει την αρχή τη προφύλαξη. Χωρί να παρατείνει την εξουσιοδότηση για αυτέ τι δραστικέ ουσίε, πριν από λίγε μήνε κάναμε συζήτηση για το θέμα αυτό μεταξύ ημών και εκπροσώπων του ΆΙΑΡΚ και τη ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ ισχυρίστηκε ότι έχουν έναν μεγάλο αριθμό, ικανό αριθμό επιστημονικών μελετών στα χέρια τους ως ε, αναφορά για την αποφασή τους. Όμως ε, και στο κοινό έχουν διαρρεύσει πάρα πολλές πληροφορίες και το κοινό είναι ενημερωμένο. Η ΆΕΡΚ δεν φαίνεται να είναι τη ίδια άποψη βεβαίω, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρατείνει την εξουσιοδότηση τη γλυφωσάτη για 15 χρόνια. Γιατί? Γιατί πρόκειται για την μέγιστη δυνατή περίοδο που θα μπορούσε να προβλέψει. Δεν μπορούσε να κάνει μια διαφορετική πρόταση, διότι τα περισσότερα μέλη του Κοινοβουλίου δεν είναι υπέρ τη παράταση τη εξουσιοδότηση, γιατί τόσα πολλά χρόνια σε κάθε περίπτωση. Και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει μια εναλλακτική πρόταση. Ξέρουμε ότι υπάρχει κίνδυνος από την ουσία αυτή για τα θηλαστικά και τους ανθρώπους. Καταστρέφει όχι μόνο τα αγριόχορτα, αλλά τους μύκητες, τα βακτηρίδια, τα αγριόχορτα και τα φύκια. Ε, είναι λοιπόν μια μεγάλη απειλή κατά της βιοπικιλότητας. Παρά τις αντιπαράθεσης λοιπόν μεταξύ της Άρη και της ΕΦΣΑ ε, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν και οι δύο. Θέλουν να ακούσουν τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου τα επιστημονικά στοιχεία της ΕΦΣΑ να διαταθούν και στο κοινό. Αλλά λέει η ΕΦΣΑ σε μία μεμονωμένη μελέτη ότι η γλυφοσάτη δεν προκαλεί γενετικά προβλήματα. Περισσότερες όμως μελέτη και μελέτες και η συστηματική έρευνα στη βιβλιογραφία δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές απειλές για τα θηλαστικά και τους ανθρώπους. Αν δούμε λοιπόν και τις καρκινογόνες ουσίες, αυτό αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Για τους ενδοκρινικούς διακαταράκτες στου στους ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή με την παράτασή τη, δεν προάγει καθόλου την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή αυτή ζώων ή το περιοριστή του περιβάλλοντο. Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντο η ευρωπαικη επιτροπη δεν αξιοποιεί τα εργαλεία που διαθέτει ή ε, δεν μπορεί να εφαρμόζει καν την αρχή τη προφύλαξης. Η ομάδα μας λοιπόν θεωρεί ότι όλα αυτά δεν συνάδουν με τα μέτρα του κανονισμού 1107 του 2009. Η ερώτησή μα λοιπόν είναι κατά να μπορείτε να αποσύρετε την πρότασή σας για παράταση μέχρι να εκπονηθεί ανεξάρτητη μελέτη για την ε, ταξινόμηση της γλυφωσάτης. Επίσης ζητούμε από την ΕΦΣΑ να ενημερώσει το κοινό να δημοσιεύσει τις επιστημονικές της πληροφορίες το ίδιο και η Γενική Διεύθυνση Σάντα πρέπει να λάβει σοβαρά την διάσταση προστασία τη υγεία των ανθρώπων. Αυτή είναι η υποχρεώσή σα. Πρόεδρο, ευχαριστώ συναδελφοί. Έχουμε περισσότερους από 20 αγορητέ. Εάν ο καθένα μιλάει για 5 λεπτά, νύχτα. Ευχαριστώ. Τώρα, ο κύριος Πεντιτσίνη, εκ μέρου τη EFTD. Ε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότερος. Ε, φαίνεται απίστευτο, αλλά και πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε με την επίκληση τη αρχή τη υποφύλαξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα προτείνει αυτή την παράταση τη χρήση τη γλυφοσάτη για άλλα 15 χρόνια. Βλέπουμε στοιχεία για την γλυφοσάτη, το βρίσκω εγώ αυτό ουσία σε 14 διαφορετικέ μάρκε απορριπαντικών και δεν είναι το πρόβλημα μόνο η υδροφόροι ορίζοντα και η βιοπικιλότητα. Είναι μια ουσία που περνάει απευθεία στην τροφική μα αλυσίδα. Κι όμω ε, η Γερμανία και η ΕΦΣΑ μα έχουν πείσει ότι η γλυφοσάτη δεν αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τον άνθρωπο. Αλλά έχουν βασιστεί σε μελέτε που χρηματοδοτούν οι ίδιε πολυεθνικέ που παράγουν προϊόντα με γλυφοσάτη. Η, ε, το Επιστημονικό Κέντρο για την Ογκολογία με την συμμετοχή εκατοντάδων εμπειρογνωμόνων από 11 χώρε βρήκε άμεση σχέση μεταξύ τη παρουσία λεμφώματο και τη γλυφοσάτη. Η γλυφοσάτη λοιπόν έχει ταξινομηθεί ω μάλλον καρκινογόνο για τον άνθρωπο, σύμφωνα με την ΕΦΣΑ. Η γλυφοσάτη δεν πρέπει να επανεξουσιοδοτηθεί, όχι μόνο γιατί ρηπαίνει, αλλά και γιατί ε, βράχει πρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Ήθελα να ξέρω λοιπόν γιατί η γλυφοσάτη περνάει ακόμα και στα δημητριακά, που ε, τα παιδιά μας μπορεί να καταναλώνουν το πρωί ε, και σε καταστάσεις ε, που η κατανάλωση γίνεται λίγη ώρα μετά τη συγκομιδή. Πώς λοιπόν μπορεί αυτή η ουσία να καταναλώνεται και τόσο ε, αμέριμνα ενώ μπορεί να είναι και καρκινογενής. Πώς δεν λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο ότι μπορεί να είναι ενδοκρινικός διταράκτης και πώς δεν λαμβάνεται υπόψη να θέτει επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε κατά τις ουσίες αυτής μεταξύ άλλων χημικών ε, ουσιών. Ρωτάω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι αρχές για να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης και αν δεν το κάνετε τώρα πότε θα το κάνετε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντορνανό, εκ μέρους της ΙΕΝΕΦ. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να διευκρινίσω ένα διαδικαστικό ζήτημα. Όλες ε, οι πολιτικές ομάδες ε, είναι υπέρ της αντίρρησης, ενώ εμείς είμαστε μόνοι μας. Η δική μας ομάδα, δεν έχει τον ίδιο στόχο, ή έχει μείνει απομονωμένη. Ε, στόχος της ομάδας μας είναι να εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των πολιτών, την υγεία, την υγεία τους και το περιβάλλον και να ξεπεράσουμε τις κομματικές αντιπαραθέσεις, χάρη αυτού του κοινού συμφέροντος. Όλοι συμφωνούμε για τα αποτελέσματα της γλυφοσάτης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται εμπορικά με τοξικές βοηθητικές ουσίες. Θα πρέπει να πάρει λίγη απόσταση από την νομοθεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να λάβει υπόψη και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή και τη μαζική χρήση των αντιβιωτικών. Αυτό είναι εποδό στα τελευταία χρόνια, ενώ η γλυφοσάτη θεωρείται αντιβιωτικό. Μάλιστα, έχουν κατατεθεί διπλώματα ευρυστεχνία για τη χρήση τη γλυφοσάτη ω αντιβιωτικού. Η καταπολέμηση τη μικροβιακή αντοχή, λοιπόν, περνάει από μια ενισχυμένη προφύλαξη ό,τι αφορά τη χρήση ουσιών που χρησιμοποιούνται ω αντιβιωτικά. Γιατί λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήγε πολύ μακριά. Θεωρούμε ότι το επιστημονικό πλαίσιο είναι ιδιάζων. Αφενός ε, ε, έχουμε διαφορά του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον καρκίνο από, την, ε, από το δικό μας Οργανισμό Ασφάλειας των Τροφίμων και η το Γερμανικό Ινστιτούτο Einrich Μπολ ε, υπεσήμανε σημαντική έκθεση των πιο ευάλωτων ομάδων στη γλυφοσάτη. Έχουμε λοιπόν δύο βασικούς λόγους για να είμαστε ε, επιφυλακτικοί και συνετοί. Επίσης, επισημάναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη να τηρήσει και να σεβαστεί την αρχή της προφύλαξης. Μάλιστα, επ' ευκαιρία μιας απόφασης που αφορά τη θέση σε εμπορία φυτοφαρμάκων, ζυζανιοκτώνων φανταζόμασταν ότι θα δείξει αυτή τη σύνεση και την προφύλαξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνει ένα νέο, μια νέα μελέτη του κινδύνου τουλάχιστον ή και ή να εφαρμόσει νέα κριτήρια και νέα προσέγγιση. Επιπλέον, η υπόσχεση της δημοσίευσης του καταλόγου βοηθητικών ουσιών που απογορεύονται λόγω του ταξικού τους χαρακτήρα δεν είναι σοβαρή πρόταση και απάδει από την αρχή της χρηστής διαχείρισης του καταλογου βοηθητικων ουσιων που απογορευονται λογω του ταξικου του χαρακτηρα δεν ειναι σοβαρη προταση και απαδει απο την αρχη της χρηστη διαχειρισης του κινδυνου και της προφύλαξης. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να προβλέψει ένα νέο στάδιο Νομοθετική μεταρρύθμιση συμπεριλαμβάνοντα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τη γλυφωσάτη, η χρηματοδότηση έρευνα και ανέβρεση λύσεων και εναλλακτικών προϊόντων θα ήταν ένα αποφασιστικό βήμα προ την κατεύθυνση αυτή. Τέλο, τα κράτη-μέλη είναι διχασμένος προ το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έπρεπε να διαθέσει χρόνο σε διαβουλεύσεις προκειμένου να επιδιώξει μία σύγκληση των κρατών μέλων. Ευχαριστώ κύριε Δεμεσμέκερ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είχα αποφασίσει να στηρίξω την αντίρρηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανανεώσει την έγκριση για την ε, γλυφοσάτη. Φαίνεται να μην υπάρχει επιστημονική συνένεση στο θέμα αυτό, σύμφωνα με την ΕΦΣΑ. Η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος ουσία, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο έχει καταλήξει ότι μάλλον πρόκειται για καρκινογόνο ουσία. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των βοηθητικών co-formulants. Αυτό αναφέρεται στα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ. Και ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για το Καρκίνο, η IARC, εξέτασε το θέμα των βοηθητικών, αλλά από διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς ε, μήλα με πορτοκάλια, να συγκρίνει μεταξύ τους διαφορετικά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται επίσης να καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Γιατί λοιπόν ε, η λιποαμίνη ως βοηθητικό να χρησιμοποιείται ως λύση αυτό αποτελεί μέρος της λύσης, όχι όμως μια συνολική λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι επέλεξε το μέγιστο διάστημα ανανέωσης, δηλαδή 15 έτη. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν περαιτέρω μελέτες πάνω στη γλυφοσάτη και τα βοηθητικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου. Η ΕΦΣΑ ήταν αντικειμενική, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί να εξετάζουμε μόνο τις δραστικές ουσίες, θα πρέπει να εξετάζουμε και τις βοηθητικές. Συμφωνώ με όσους θέλουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά ε, ε, τις ε, ενδοκρινολογικές διαταραχές. Νομίζω ότι υπάρχουν υπορβολικά πολλές ανησυχίες για να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό στηρίζω την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Παύλ Πότς τον ε, συνεισηγητή που είπε ότι δυστυχώς ε, είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες επί της ουσίας εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος μπορεί να επιστήσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένας ε, λόγος παραπάνω λοιπόν να υψώσουμε και μάλιστα στεντόρια τη φωνή μας σε ένα βήμα. Επανειλημμένα ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που εγκύπτουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και εγώ συνυπέγραψα το ψήφισμα, μάλιστα όχι εκ μέρους ομάδας, αλλά προσωπικά, γιατί η ομάδα μου δυστυχώς εξακολουθεί να είναι διχασμένη στο ζήτημα αυτό. Θα σας δώσω τους ε, λόγους, αν και το έχω κάνει επαρελειμμένος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει στην περίπτωση αυτή ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε να κάνει για το ζήτημα αυτό. Ε, στο θέμα της ανανέωσης ή όχι της άδειας για τη χλυφοσάτη. Φαίνεται, φάνηκε μεροληπτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έπρεπε αμερόληπτα να κρίνει με βάση επιστημονικά κριτήρια ε, τα θέματα αυτά που έχουν πολιτικές ε, διαστάσεις, επιστημονικές διαστάσεις, αλλά και μια ιδιαίτερη απήχηση στην κοινή γνώμη. Μάλιστα, το Διεθνέ Κέντρο έρευνα του Καρκίνου τη ΠΟΗ μα λέει ότι ενδέχεται να είναι καρκινογόνος η γλυφοσάτη, ενώ οι εμπειρογνώμονε ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ασφάλεια των Τροφίμων λέει όχι αποκλείεται. Δεν είναι η πρώτη φορά τέτοιων αντικρουόμενων επιστημονικών ε, πορισμάτων. Δεν συμφωνούν οι εμπειρογνώμονε. Ε, έχουν υπόνοιε, αλλά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία επιφύλαξη. Είναι κατηγορηματική υπέρ τη ανανέωση. Ενώ η, δεν είναι μόνο η δραστική ουσία γλυφοσάτη που είναι προβληματική, αλλά και η προσθήκη του κοκτέιλ αυτών των βοηθητικών ουσιών που απαρτίζουν αυτό το ζυζανιοκτόνο, το Roundup και το καθιστούν ε, καρκινογόνο, αυτό είναι προβληματικό. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε και τη χρήση του ΣΥΠΕΟΤΕΛΟ αμήν, εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλαξης, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή από τους 500 βοηθητικές ουσίες μόνο αυτό, αυτή την ουσία θα απαγορεύσουμε. Αυτό εννοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προφύλαξη, αρχή της προφύλαξης, απαγορεύοντας μόνο ένα από τα 500 που είναι επικίνδυνα. Επίσης, ε, δεν είναι κάθε μέρα που βλέπουμε, όπως το θέμα αυτό, μια Προεδρία που έρχεται σε αντιπαράθεση και δημόσια μάλιστα αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν είναι μόνο της η Ολλανδική Προεδρία εδώ. Πέντε κράτη-μέλη είναι κατά της πρώτης ανανέωσης προς το παρόν. Στο μέλλον ελπίζω να συμπαραταχθούν με τη θέση αυτή και άλλα κράτη-μέλη. Και 243 εκατομμύρια πολίτες. Ελπίζω στις αρχές Μαρτίου ε, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ε, κατάλαβε ακριβώ ε, ότι δεν θα είχε ενισχυμένη πλειοψηφία και αποφάσισε αναβολή μέχρι το Μάιο. Φαντάζομαι αυτό ήταν το σκεπτικό τη Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, τη μόνιμη Επιτροπή. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι χαμένη από χέρι αυτή η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να επανεξεταστεί. Έχουμε δύο ψηφίσματα εδώ για συζήτηση και θα ζητούν κάπως αφελώς αμέσως να απαγορεύσουμε τη γλυφοσάτη. Αυτό καταλάβατε. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο των ψηφισμάτων. Ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το καθήκον τη, να αποσύρει την πρόταση και να καταθέσει νέα. Δεν θα υποκατασταθούμε εμεί στο έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητούμε ένα χρονοδιάγραμμα, σταδιακή απαγόρευση, ένα κατάλογο των προβληματικών βοηθητικών ουσιών και όχι μόνο μία βοηθητικής ουσίας. Επίσης να ακούσει εμά, τους εμπειρογνώμονε τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, του Γερμανού εμπειρογνώμονε, του Γάλλους εμπειρογνώμονε, την κοινή γνώμη, να μην κοφεύει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ζητούμε, όχι απαγόρευση από αύριο και όλα τη γλυφωσάτη. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμη να φέρουμε στα συγκαλά της την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, και να μην είναι τόσο ριζοσπαστική σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ο κύριος Γιάρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, για λόγους υγείας ε, δεν μπορούσε να ε, είναι παρούσα η συνάδελφος Ελά και γι' αυτό μου ζήτησε να πάρω το λόγο στο όνομά της. Παρακαλώ τους ε, συναδέρφους ε, να σκεφτούν. Πάντα λέμε ότι θέλουμε ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα μπορείτε να έχετε ό,τι αποτέλεσμα θέλετε. Και μάλιστα επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες. Και δεν θυμώνω τόσο πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο με το Συμβούλιο που με αποχή ψήφου μπλοκάρει τόσα θέματα. Η ΕΦΣΑ ανέθεσε στο Γερμανικό Ινστιτούτο Αξιολόγησης ε, Κινδύνου ε, την ε, σχετική μελέτη. Η Γερμανία όμως απέχει από την ψηφοφορία. Δηλαδή η Γερμανία δεν στηρίζει το αποτέλεσμα του δικού της Ινστιτούτου. Εμένα αυτό με κάνει να σκέφτομαι διάφορα. Ένα παράδειγμα να σας δώσω που με βάζει σε σκέψεις. Διαπιστώνεται ότι στα ούρα υπάρχουν κατάλοιπα γλυφοσάτης που είναι πιο ψηλά από τα, τις οριακές τιμές για το πόσιμο νερό. Το να Συγκρίνουμε όμως το πόσιμο νερό με τα ούρα ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος. Σας παρακαλώ λοιπόν να είμαστε απολύτω αντικειμενικοί στη συζήτηση αυτή και σε ό,τι κάνουμε να σκεφτούμε και τις πρακτικές συνέπειες. Ε, θα πρέπει να βρούμε μία λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Οι συνάδελφοι λένε ότι ε, δεν υπάρχει πρόβλημα να απαγορεύσουμε μια ουσία, θα βρεθεί μια καινούρια. Αλλά η επόμενη ουσία που θα την αντικαταστήσει όχι μόνο θα είναι πιο δαπανήρη, αλλά συχνά έχει ακόμα χειρότερες συνέπειες για το περιβάλλον. Παρακαλώ λοιπόν να το σκεφτείτε αυτό. Εκ μέρους ε, λοιπόν της συναδέλφου Τελάη ζητούμε αντικειμενική συζήτηση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να απαγορεύσουμε στο Συμβούλιο σε πολλές περιπτώσεις να απέχει από την ψηφοφορία. Θα πρέπει ε, να δηλώνει τι θέλει, ναι ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία για τα γλυκοσάτη. Κάποιες από τις ανησυχίες τις καταλαβαίνω, κάποιες άλλες λιγότερο. Αλλά αυτό που θέλω να πω οπωσδήποτε είναι ότι αναγνωρίζω την πραγματική ανησυχία, τη βαθιά ανησυχία του κυρίου Πότς και έχει αναπτύξει πολύ σωστά τα επιχειρήματά του. Νομίζω ότι κάποιοι από τους υποστηρικτές της αντίρρησης ε, έχουν αναπτύξει τα επιχειρήματά τους εδώ που ουσιαστικά προσβάλλουν το σκοπό μας, αλλά το είπα, τι να κάνουμε, συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ε, Ανησυχώ κάπως για το ψήφισμα, γιατί θεωρώ ότι είναι ανακριβές σε πολλά σημεία. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι κακώ η ομάδα μου θεωρεί ότι πρέπει να εξετάσουν κάποια από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γλυφοσάτη, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω ότι η ΕΦΣΑ έχει χάσει την αξιοπιστία τη και ε, ε, δεν θα πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά την ΕΦΣΑ. Δεν θυμάμαι να το λέει κανεί αυτό σε αυτή την αίθουσα, ιδίω τη φορά που ήρθε η ΕΦΣΑ για να κάνει τη δήλωσή τη. Φαίνεται ότι είχε μια διαφορετική άποψη με τι απόψει που ακούγονταν εδώ στην αίθουσα, παρόλο που ήταν αντίθετη με, άλλες επιστημονικά, με, με άλλα επιστημονικά πορίσματα. Τώρα κάποιοι δεν, διαφων, δεν συμφωνούν πια με την ΕΦΣΑ και θέτουν να αμφιβόλο την αξιοπιστία του. Ε, δεν είναι έτσι. Η ΕΦΣΑ έχει τη δική τη τη δουλειά να κάνει, έχει κάποιε αρμοδιότητε, εξέτασε την ουσία και κατέληξε σε πορίσματα. Εδώ λοιπόν εξετάζουμε διαφορετικά πράγματα τελείω μεταξύ του ε, ε, όταν μιλάμε για τον IARC και την ΕΦΣΑ. Ε, ο IARC κοιτάζει τι χημικέ ουσίες και τις φόρμουλές τους, όχι τα ίδια με την ασφάλεια που κοιτάζει η ΕΦΣΑ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μας είπε η ΕΦΣΑ και να αποφασίσουμε αν θέλουμε να τα υποστηρίξουμε ή όχι. Και ακριβώ επειδή νομίζω ότι εδώ ξεπερνάμε λίγο τώρα τι επιχειρηματολογίε μα, δεν μπορώ να στηρίξω το, την αντίρρηση. Κυρίω γιατί ο κανονισμό φαίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την προστασία τη υγεία των ανθρώπων και των φυτών. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ούτε ισχύει ότι δεν καταφέρνει να εφαρμόσει την αρχή τη προφύλαξη. Η αρχή τη προφύλαξη δεν είναι μια απλουστευτική έννοια. Εάν υπάρχει κίνδυνο να συμβεί κάτι, δεν σημαίνει ότι το απαγορεύει. Είναι μια ε, εξέταση του θέματο με έναν τρόπο που προσπαθεί να βρει το σωστό σημείο ισορροπία. Αυτή είναι η αρχή τη προφύλαξη. Εδώ λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει να λέμε ότι ουσιαστικά εμποδίζει τη λειτουργία του κανονισμού. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν όσοι προτείνουν αυτή την αντίρρηση είναι να παρακάμψουν την κανονική την διαδικασία, η οποία λέει ότι είναι εφαρμοστική πράξη στην οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν εμπειρογνώμονε. Οι εμπειρογνώμονε αυτοί δεν έχουν ακόμη αποφανθεί, δεν έχουν τοποθετηθεί δημοσίω. Ξέρουμε ότι συζητούν, ότι διαπραγματεύονται, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Οπότε, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει του εφαρμοστικού κανονισμού και νομίζω ότι έτσι όπω έχει συνταχθεί το κομμάτι αυτό είναι παράλογο και διαβάσιμο. Επίση, καλείται η Επιτροπή να μην προβλέψει την παράταση τη γλυφοσάτη με ένα διαφορετικό και σαφέ χρονοδιάγραμμα. Μα υπάρχει και το είπαν. Είπαν ότι θα το προτείνουν μέχρι τον Ιούλιο ε, και θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ε, υποκατάσταση τη γλυφοσάτη. Επίση, στο σημείο 4 καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά κάποιος ε, φέρνει αντιρρήσεις για το χρόνο της ομιλίας σας. Μας συγχωρείτε. Α, ευχαριστώ. Καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ανεξάρτητη μελέτη για την κατηγοριοποίηση της γλυφωσάτης. Μα αυτό γίνεται ήδη. Δεν καταλαβαίνω πόσοι άνθρωποι που ε, υπέγραψαν αυτό το ψήφισμα το διάβασαν κιόλα. Στο 5 καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαλύψει όλα τα επιστημονικά στοιχεία. Ζήτω! Με αυτό συμφωνώ κι εγώ. Θα έπρεπε. Ναι. Αλλά δυστυχώ το σημείο αυτό το συνοδεύουν και όλα τα υπόλοιπα. Στο 6 καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει εντολή στον ε, ΦΑΟ. Με ποιο επίπεδο ασφάλεια που θα πρέπει να το μελετήσουν. Και αυτό αν δεν έχουμε ήδη μελετήσει του ενεργού ουσίε που θέλουμε να ερευνηθούν. Δεν συμφωνώ λοιπόν με όλα αυτά. Θα ήθελα να ε, διατυπωθούν με τρόπο λογικό διότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να θέσουμε κάποιες απορίες στην ΕΦΣΑ, αλλά εδώ έχουμε αρχίσει να γινόμαστε ιστηρικοί και να ξεπερνούμε τα όρια. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κουτέμα για την Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι στην ομάδα των φιλελευθέρων συζητήσαμε το απόγευμα αυτό το θέμα, αλλά δεν έχουμε αποκριστελωμένη ή ρητή γνώμη κατά της ανανέωσης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιστημονικές γνωματεύσεις και επιστημονικά πορίσματα. Δεν θα πρέπει να πολιτικοποιήσουμε τη συζήτηση ή να είμαστε επιλεκτικοί στα επιχειρήματα. Η Επιτροπή... Ζητήσαμε οι φιλελεύθεροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ειμαστε επιλεκτικοι στα επιχειρηματα η επιστημονικές έρευνες για να στοιχειοθετήσει την πρότασή της. Επίσης, η απαγόρευση της γλυφοσάτης μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα, γιατί η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος χρήστης της γλυφοσάτης και φυσικά οι γεωργοί έχουν επίγνωση των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει μια πιθανή απαγόρευση της ουσίας αυτής. Βέβαια και οι συμπολίτες μας ανησυχούν, γιατί όλο και περισσότεροι γεωργοί ε, και κυπουροί εφαρμόζουν την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση των, ε, για τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Τι σημαίνει τώρα ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σημαίνει χρήση φυτοφαρμάκων και ζανιοκτώνων με υπεύθυνο τρόπο και μόνο όπου δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις ή μέθοδοι. Και υπάρχουν τρόποι για να μειώσουμε σημαντικά τη χρήση φυτοφαρμάκων και ζυζανιοκτώνων. Αυτό θα πρέπει να διερευνήσουμε. Και όχι απλώς ε, να απαγορεύσουμε κάποια ζυζανιοκτώνα ή φυτοφάρμακα. Γιατί οι γεωργοί και οι κυπουροί θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσουν ε, τις ε, καλλιεργίες τους, να έχουν ένα δίκτυο ασφαλείας. Βέβαια, να καταφεύγουν πρώτα σε εναλλακτικέ πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, αλλά να έχουν ε, ως έσχατη λύση και ένα ζανιοκτόνο. Για παράδειγμα, το ξεχέρσωμα, ε, η καύση των ζυζανίων με τη χρήση φυσικών τοξινών είναι μια λύση πολύ λιγότερο επιζήμια για το περιβάλλον, πολύ πιο φιλοπεριβαλλοντική. Επίσης, να λάβουμε υπόψη και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο μιας πιθανής απαγόρευσης ε, της γλυφοσάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι τρίτες χώρες δεν θα στενιστούν την απαγόρευση και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή τη δραστική ουσία, κάτι που θα δημιουργήσει τον ανταγωνισμό εις βάρος των γεωργών μας και της επιστηστικής βιομηχανίας μας. Ευχαριστώ κύριε Σλίζε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο και επίμαχο το θέμα. Νομίζω όμως ότι όλοι συμφωνούμε στο εξής και θα ήθελα να το τονίσω παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Η Κομισιόν πρότεινε να απαγορευτεί η να απαγορευτούν οι λιποαμίνες, τα λοαμίν, και ήδη το 2012 Είχα απευθυνθεί στους ε, επιτρόπους Σεντάλη και Ποτόφνικ και νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό. Κατά τα άλλα είναι δύσκολο το θέμα και νομίζω ότι κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δώσει τη λαθασμένη εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την γλυφοσάτη. Εγώ ε, ως γιατρός ε, νομίζω πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να ε, την καταναλώνουμε σαν το νερό. Είναι προβληματική η ουσία. Αλλά θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε το θέμα της απαγόρευσης, διότι ακόμα και η βαθμιαία απαγόρευση, ένα phasing out, θα οδηγήσει σε χρήση εναλλακτικών μεθόδων για τις οποίες ε, έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες για να γνωρίζουμε ε, αν ε, είναι τελείως απειλαγμένες από προβλήματα. Και με εισαγωγές δεν θα έχουμε βελτίωση τελικά. Θα έχουμε και συνθήκες ανισού ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Ελπίζω όμως ε, στον δρόμο μας προς την Ολομέλεια να μπορέσουμε να έχουμε ε, επικοδομητικές συμβιβαστικές προτάσεις. Αύριο έχουμε την πρώτη ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ε, ξεκαθαρίσουμε το θέμα των βοηθητικών ουσιών και μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε συμβιβαστική πρόταση σχετικά με τις διάφορες εφαρμογές ε, της γλυφοσάτης. Ε, ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε πιο αναλυτική συζήτηση, διότι με ένα απλό ναι ή όχι δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε σωστά το πολύπλοκο αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο. Γκρότε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα αν θα πρέπει να ψηφίσουμε ναι, όχι, αποχή. Αυτά είναι μάλλον λαϊκιστικές ε, μέθοδοι. και ε, αν ε, τα κράτη-μέλη δεν ε, συμμετέχουν στις ψηφοφορίες, νομίζω ότι μάλλον καταλήγουμε σε τελείως διαφορετική νοοτροπία. Πάντως είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Θα ήθελα να πω ότι πέρα από την αντικειμενική συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΦΣΑ δεν έχουν εφερθεί πολύ σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περνάει πολύ δύσκολες εποχές και δεν ότι έχει πολύ νόημα η επιχειρηματολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στο θέμα αυτό. Έχουμε μελέτη της ΕΦΣΑ αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν και τα τελικά προϊόντα σε σχέση με τη γλυφοσάτη. Το κοινοβούλιο μας έχει καθήκον να εξετάζει τις προτάσεις και όχι απλά να υπερψηφίζει τις προτάσεις ε, ο Διεθνής ε, Οργανισμός ε, για την Υγεία αναφέρθηκε στα κατάλοιπα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μελέτες που να δείχνουν ό,τι αποτέλεσμα θέλουμε. Νομίζω ότι, η... ότι θα πρέπει να προσέξουμε τη διαδικασία. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να προσέξει πολύ στο μέλλον και να αλλάξει τις διαδικασίες και τις ΕΦΣΑ. Νομίζω ότι καλά θα κάνουμε λοιπόν ε, να εισάγουμε ε, νέες ε, μεθόδους εργασίας στο θέμα αυτό. Το θέμα δηλαδή δεν είναι αν αύριο θα ψηφίσουμε ναι ή όχι, το θέμα είναι η όλη διαδικασία. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε την αντίρρηση. Ο κύριος Φαρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ο προλαλής σας του ΕΛΚ, πρέπει να γίνει συζήτηση. Μια σοβαρή συζήτηση για να λάβουμε αντικειμενική απόφαση. Αυτό ακριβώς μας λείπει. Στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα περιπλοκό και το οποίο προκαλεί διαφωνίες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ίδιων των επιστημόνων και μεταξύ των απόψεων των κρατών μελών. Η ΕΦΣΑ από τη μια θεωρεί την δραστική ουσία της γλυφωσάτης ε, ως από τις χειρότερες, ενώ η θεωρεί τη δραστική ουσία της γλυφοσάτης και την ε, τοποθετεί σε μια άλλη κατηγορία, με τους συνμορφωτές, με τις βοηθητικές συγγνώμη ουσίες. Θεωρεί η ΕΦΣΑ ότι η ουσία δεν είναι καρκινογενής, ενώ... Ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί το προϊόν αυτό καρκινογενές. Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι αποκλίνουν μεταξύ τους. Είναι διαφορετικά. Η, όλη αυτή η μελέτη, η ευρύτερη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που κατέληξε στο πόρασμα ότι η γλυφοσάτη είναι καρκινογόνος, ε, θέλω να ξέρω πώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εμεί δεν είμαστε ούτε επιστήμονε, είμαστε πολιτικοί, άντρε και γυναίκε, και η πρώτη μα υποχρέωση είναι να προσπιζόμαστε την δημόσια υγεία τι πρέπει να θεωρήσουμε ότι ισχύει. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι όσο έχουμε επιτάπητος δεν αρκούν για να επιτρέπουν την ε, χρήση της ουσίας αυτής ε, χωρίς πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης που προβλέπει την μη συνέχιση της χρήσης της ουσίας αυτής μέχρι να υπάρχουν πιο διεξοδικά και πιο πιστικά επιστημονικά στοιχεία. Ε, ήθελα να πω επίσης ότι Τελικά έχουμε μεγαλύτερη σύγχυση σήμερα για το θέμα αυτό ε, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από μερικού μήνε και αυτό εξαιτία ακριβώ τη τοποθέτηση των ε, διαφόρων επιστημόνων που διαφωνούν μεταξύ του και θέλετε να αποκλίνουν στι απόψει του. Είμαστε λοιπόν πιο μπερδεμένοι από ό,τι στην αρχή. Ο κύριο Πότ είπε, το είπε στην αρχή προηγουμένω, ότι έχουμε μια μελέτη που ιδιαίτερα διεξοδική για την παράταση τη ε, εξοδότηση τη χρήση τη ουσία αυτή. Συμφωνώ 100% μαζί σα αλλά μιλάμε για μία ουσία, για, την παράταση χρήση μια ουσία για πάνω από 15 χρόνια που μπορεί ενδεχομένω να είναι εν μάλλον ε, απειλή για τη δημόσια υγεία. Δική μας λοιπόν υποχρέωση είναι να επιλέξουμε την ε, βέλτιστη λύση για την δημόσια υγεία μέχρι να γίνει μια πιο τεκμηριωμένη μελέτη από την επιστημονική κοινότητα με στοιχεία τα οποία να μας οδηγήσουν σε κάποιο τελικό συμπέρασμα και αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε αυτά τα χειροπιαστά στοιχεία που να μας επιτρέπουν να αποφασίσουμε με τρόπο σαφή και ήσυχη τη συνείδησή μας ε, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν δεν είμαι σε θέση να αποφασίσω και δεν μπορώ να εγκρίνω την εξουσιοδότηση της παράτασης, την παράταση μάλλον της εξουσιοδότησης χρήσης της ουσίας Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Χόισλινγκ. Ναι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη που με την αποχή τους σταμάτησαν τη διαδικασία αυτή, διότι αυτό που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανέναν περιορισμό δηλαδή ε, στην χρήση και έγκριση για 15 χρόνια, Δεδομένου ότι εδώ και δύο χρόνια συζητάμε πολύ επικριτικά το θέμα, αποτελεί σκάνδαλο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει καν κάτι τέτοιο. Το να μην υπάρχει καν περιορισμός στην χρήση σημαίνει τι. Σημαίνει ότι ο κάθε γεωργός ε, την εβδομάδα πριν την συγκομιδή μπορεί να ψεκάσει τα, ε, τα ε, φυτά, τα δημητριακά και μετά να τα πουλήσει σε ε, αρτοποιία. Αυτό είναι ένα παράδοξο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας το οποίο δεν θα το πίστευε κανείς. Επίσης το να ψεκάζει κανείς αυτή την ουσία στον κήπο του και αυτό είναι απαράδεκτο. Σκεφτείτε τι επιτρέπεται. Γιατί, γιατί να πρέπει να εξαντλήσει κανείς ε, την ε, μέγιστη περίοδο έγκρισης της 15 ετίας. Ευχαριστώ λοιπόν τα κράτη-μέλη που τουλάχιστον μπλόκαραν τη διαδικασία. Λαμβάνουμε τόσες αντιδράσεις από ε, πολίτες που ανησυχούν για το θέμα αυτό που νομίζω ότι αποτελεί ε, δικαίωμά μας ως ευρωβουλευτές να ε, Υποβάλλουμε την αντίρρηση αυτή. Πολλές μελέτες για την βιοπικιλότητα μας δείχνουν ότι η βιοπικιλότητα μειώνεται κατά 40% στις ε, περιοχές, στις εκτάσεις όπου χρησιμοποιείται η γλυφοσάτη. Δεν μπορούμε λοιπόν να αιτιολογήσουμε πια την χρήση αυτής της ουσίας. Ούτε αληθεύει ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση στη χρήση της γλυφοσάτης. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, ε, γεωργοί βιολογικών καλλιεργιών αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι ε, δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ουσίας αυτής. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται επειδή είναι οικονομική, για οικονομικούς λόγους όχι επειδή προστατεύει η ουσία αυτή το περιβάλλον ή επειδή ε, μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την ε, αλλαγή του κλίματος. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση της ουσίας αυτής, για καθαρά οικονομικούς λόγους χρησιμοποιείται. Και όποιος ε, δεν μπορεί να καλλιεργήσει ε, τρόφιμα χωρίς τη γλυφοσάτη, μήπως να ξανασκεφτεί το επαγγελμά του. Υπάρχουν εναλλακτικές. Γι' αυτό επιμένω στο θέμα αυτό. Εάν δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, να εμποδίσουμε την έγκριση, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει περιορισμός στη χρήση. Σίγουρα χρειαζόμαστε περιορισμό στη χρήση του ουσίας. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τη διαδικασία. Αυτή η αδιαφανής διαδικασία θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν. Υπάρχουν ε, ε, ε, δημόσια διαθέσιμες σε μελέτες, ενώ δεν, είναι, δεν έχει δημοσιευτεί αυτή τη ΣΕΦΣΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έχω να πω λίγα λόγια. Ας μην ξεχνούμε, ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι είχαμε μια πρώτη νίκη εις βάρος Μονσάντο που μας δηλητηριάζει εδώ και μια τριαντακονταετία με το ζανιοκτόνο του το Roundup που περιέχει γλυφοζάτη. Είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε, να θυμίζουμε αυτή τη νίκη και να κατονομάζουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τη Μονσάντο. Πρόκειται για μια εταιρεία που χρόνια ολόκληρα και εδώ και παντού στον κόσμο κάνει ε, εντατικότατο λόμπινγκ και έχει ένα και μόνο στόχο και φιλοδοξία αποκλειστικά, το κέρδος. Και ας μην ξεχνούμε ότι όταν επιτιθέμεθα σε αυτό το ζενιοκτόνο, το Roundup, και είμαστε κατά της γλυφοσάτης, ε, χτυπούμε τη ρίζα και τον γερεσιουργό λόγω ύπαρξη ε, τη Μονσάντο. Γιατί το Roundup, αυτό το ζωνιοκτόνο, αντιπροσωπεύει το 40% του ετήσιου τζίρου τη εταιρεία Μονσάντο. Και όταν έχουμε ένα τέτοιο θέμα, ε, πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που δεν είναι πολιτικές, ούτε καν δεοντολογικές ε, ή δεν συνάδουν με το ήθος του Ευρωβουλευτή αλλά που μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, χρηματοοικονομικά και άλλα. Ακριβώ επειδή πίσω από όλα αυτά, πίσω μας μερικές φορές βρίσκεται αυτή η εταιρεία, η Monsanto. Και πέραν των όσων ακούσαμε από τους συναδέλφους για τους κινδύνους που διατρέχουμε, αθελά μας εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του φυτοφαρμάκου, 650.000 ε, τόνοι γλυφοσάτης ε, καταναλώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Πέρα λοιπόν αυτής της διαπίστωσης και αυτής και της ιατρικής διάγνωσης, όπως μας είπε πριν από λίγο ο δόκτωρ Πίτερ Λίζε, και ενώ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας λέει ότι πρόκειται για καρκινογόνο ουσία, εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Τροφίμων, λένε όχι, τίποτα, καμία σχέση. Και μάλιστα έχουν και μία μελέτη οι επιστημονικές γνωματεύσεις ε, που χρηματοδοτούνται από την ε, ε, αγροχημική βιομηχανία, ας μην το ξεχνούμε αυτό, και 73 εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη είναι άγνωστοι. Δεν είναι επώνυμοι και οποιαδήποτε ε, σχέση τους ε, με τη βιομηχανία δεν αποκλείεται. Αυτό το έργο λοιπόν έχουμε να κάνουμε τώρα, κυρίως το πολιτικό και να καταγγείλουμε αυτά τα θέματα και να μην ε, ντραπούμε να τα καταγγείλουμε γιατί η ουσία αυτή μπορεί να έχει ιατρικές συνέπειες δυσμενείς για την υγεία των Ευρωπαίων. Γι' αυτό και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που κατέθεσαν αυτή την αντίρρηση και εγώ θα την υπερψηφίσω. Σας ευχαριστώ κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρον παρακολουθώ τη συζήτηση αυτή. Ε, επί πολλά χρόνια ε, είμαι γεωργός. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχω χρησιμοποιήσει γλυφοσάτη ούτε το round-up, ούτε τα επόμενα 20 χρόνια σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο. Ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω τη συζήτηση που διεξάγεται εδώ. Δεν έχω επαφές με την Μονσάντο και αυτό θα ήθελα να το πω. Επί 40 χρόνια δεν είχαμε τέτοια συζήτηση σχετικά με την τοξικότητα της γλυφοσάτης. Από πού ήρθε ξαφνικά αυτή η συζήτηση στο παρελθόν. Έχω δει παρόμοιες περιπτώσεις. Η ατραξίνη χρησιμοποιεί όταν επί 30 χρόνια δεν υπήρχε συζήτηση και η συζήτηση ξεκίνησε όταν ε, ε, εξέπνευσε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, της συγκεκριμένης εταιρείας. Ε, επειδή μειώθηκε η τιμή του προϊόντος, η εταιρεία ήθελε ε, να σταματήσει η κατανάλωση του προϊόντος αυτού. Μήπως λοιπόν η Μονσάντο βρίσκεται πίσω από αυτήν την κίνηση για να μπορέσει να μας πουλήσει πιο ακριβό προϊόν. Δεν θέλω να κατακρίνω την ΕΦΣΑ, αλλά και στη Γερμανία υπάρχει ε, Γερμανικό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση Κινδύνου. Και ε, σε πρόσφατη του συνέντευξη ο πρόεδρος του Ινστιτούτου είπε ότι η γλυφοσάτη έχει την ίδια, ε, την ίδια επικινδυνότητα με το αλάτι ε, όσον αφορά τις επικίνδυνες ποσότητες Το 1900 το προσδόκιμο ζωή ε, στην ε, Γερμανία ήταν 38 χρόνια παρότι δεν χρησιμοποιόταν καμιά ε, χημική ουσία. και τώρα μιλάμε κάθε φορά που αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής κατά τρεις μήνες. Και όσον αφορά τις οριακές τιμές για την μπύρα, ξέρετε ότι βαβαρός είμαι. Είναι λοιπόν περίεργο που ακριβώς την ημέρα που, υπήρχε, που γινόταν η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούστηκε αυτό το θέμα. Και ο πρόεδρος Χέντελ του Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση Κινδύνου στη Γερμανία λέει ότι επικίνδυνη δόση προσλαμβάνει κανείς εάν πίνει χίλια λίτρα μπύρα την ημέρα. Νομίζω ότι η μπύρα που θα καταναλώνει κανεί, θα είναι πιο επικίνδυνη από τη δόση γλυφοσάτης. Επίσης, ο πρόεδρος Χένσελ του Ινστιτούτου αναρωτήθηκε ε, γιατί ε, ανησυχούμε για την γλυφοσάτη στα ούρα. Επικίνδυνο θα ήταν αν δεν τη βρίσκαμε στα ούρα, διότι θα σήμαινε ότι ο οργανισμός ε, δεν μπορεί να αποβάλει την ουσία. Μπορεί να συζητήσει κανείς ε, αν ε, θα ε, παρατείνουμε την έγκριση για 10 ή 15 χρόνια, αλλά υπάρχουν και επικίνδυνες ουσίες στη βιολογική γεωργία, όπως είναι... Ο θηλυκός χαλκός. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, έχουν ξεκινήσει την κίνηση αυτή, αλλά θα αφήσουμε τώρα αυτού να αποφασίζουν τι θα κάνουμε αντί να λέμε εμεί τη δική μα γνώμη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέλιορε. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα υπερψηφίσω το ψήφισμα διότι πιστεύω ότι πρέπει να τηρούμε την αρχή της προφύλαξης στην Ευρώπη. Υπάρχουν ανησυχίες, έχουν ε, ε, παρουσιαστεί από διάφορες πλευρές. Θα πρέπει λοιπόν να τις αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά την Μονσάντο θα ήθελα να πω ότι η Μονσάντο ε, δεν ε, παράγει μόνο τη γλυφοσάτη αλλά και τα φυτά που αντέχουν στην γλυφοσάτη και εκεί αρχίζουν ε, οι ανησυχίες μας διότι έτσι περιορίζουμε σημαντικά τη βιοπικιλότητα για να το πω με ίδιο τρόπο κιόλας. Στην Ευρώπη με την οτροφία μας, εισάγοντας τις ζωοτροφές από τρίτες χώρες, χρησιμοποιούμε προϊόντα με γλυφοσάτη και δεχόμαστε τις βλάβες που υφίστανται άνθρωποι. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης τι διαδικασία θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε εδώ, διότι δεν μπορεί η Βραζιλία και η Αργεντινή να κάνουν ακριβώς αυτό που εμείς δεν θέλουμε να έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιρπηρίκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το συζητούμε και στις κατοχώρες. Τώρα για τα επιστημονικά στοιχεία μένονται οι συζητήσει και ο Υπουργό Βαντάμ είπε και στου ελιστέ ότι γίνεται σφοδρή συζήτηση. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία και την κυπουρική, γιατί η Γεωργία χρησιμοποιούσε γλυφοσάτη εδώ και πολλά χρόνια και φάνηκε ότι σε κανονική χρήση, σε μη υπερβολική χρήση είναι ασφαλή ουσία. Με προβληματίζει αυτό το θέμα γιατί φυσικά χρειαζόμαστε τρόφιμα αλλά μας ενδιαφέρει και η υγεία και ο Επίτροπος, ο Αρμόδιος για την Υγεία, μας μίλησε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Γεωργίας και μας είπε ότι θα τα ζυγίσουν όλα, θα τα σταθμίσουν όλα και θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη και στην ΕΦΣΑ. Είπε ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΦΣΑ που έχει συμβουλευτικό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δράση με βάση τις συστάσεις και τα πορίσματα της ΕΦΣΑ. Το είπε ξεκάθαρα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τη γεωργία, την ασφάλεια και την επιστήμη. Τι να πρωτοδεχτούμε. Εμένα με έπεισε την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Ανδριοκάητες. 15 χρόνια βέβαια είναι πολύ παρατεταμένη περίοδος. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιευθούν. Αυτό είναι σημαντικό διαφάνεια. Η κυρία Σχάλτε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέρφους που πρότειναν να υποβάλουμε αυτή την αντίρρηση για την παράταση έγκρισης ε, της γλυφοσάτης. Και μόνο το γεγονός ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγεία και η ΕΦΣΑ έχουν τόσο διαφορετική αξιολόγηση της ουσία ε, θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε περισσότερες σκέψεις ε, σχετικά με το αν θα πρέπει να δεχτούμε την έγκριση αυτή ή όχι. Καταλαβαίνω ότι οι δύο αυτοί οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικέ μεθόδου για την αξιολόγηση των ε, ουσιών. Ε, η ΕΦΣΑ εξετάζει δραστικέ ουσίε, ενώ ο ΠΟΗ ε, εξετάζει τη συνέπεια στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, αν υπάρχουν τέτοιε διαφωνίε μεταξύ εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να ανησυχήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε την ουσία. Συμφωνώ λοιπόν με την αντίρρηση και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα και ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να δοθεί 15 ετή παράταση για ουσία για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι καρκινογόνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ προβληματίζομαι και ανησυχώ ιδιαίτερα, όπως και πολλοί προλαλήσαντες. Ε, οι επιδημιολογικές μεταναλύσεις ε, εργαζομένων που χρησιμοποιούσαν γλυφοσάτη έδειξε τα τελευταία 14 χρόνια ε, αυξημένο κίνδυνο για λέμφωμα. Και μάλιστα διπλάσιο ήταν ο κίνδυνος ε, για τους εργαζόμενους αυτούς που χρησιμοποιούσαν ε, ή χειρίζονταν γλυφοσάτη σε σχέση με το μέσο πληθυσμό. Έχουμε λοιπόν διάφορα στοιχεία και πολλές επιστημονικές μελέτες. Επίσης, ε, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο το 2015 ταξινόμησε τη γλυφοσάτη τις ουσίες που είναι δυνάμει καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Και ένα Ινστιτούτο από την Καλιφόρνια ε, έκρινε ότι ε, θα πρέπει να, να συμπεριληφθεί η γλυφοσάτη στις ε, καρκινογόνες ουσίες. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να εφαρμόσουμε πάνω απ' όλα την αρχή της ίνης και της προφύλαξης. Θα πρέπει να στηριζόμαστε σε επιστημονικά πορίσματα και γνωματεύσει, αλλά να λάβουμε υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντο και την δημόσια υγεία. Και πάνω απ' όλα να εφαρμόσουμε την αρχή τη προφύλαξης. Γι' αυτό και με ευνηδίασε η πρόσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση κατά 15 χρόνια τη ε, χρήση τη γλυφωσάτη. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη όλα τα επιχειρήματα που εξέθεσαν και οι και όπω σας ανέφερα και εγώ. Ε, μάλιστα οι μεταβολικές ε, οδοί όλων αυτών των ε, τοξικών ουσιών δεν έχουν διερευνηθεί δεόντως και είναι πολύ πιθανό να, να προκαλούν πολύ πιο επιζήμιες συνέπειες από ό,τι φανταζόμαστε γιατί η αρρώστια εμφανίζεται μετά από πολλά χρόνια. Οπότε Γι' αυτό ακριβώ, επειδή υπάρχουν υποψίε για την επικίνδυνοτητα τη ουσία, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνετοί και, ε, επιφυλακτικοί. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί που έχουν πρωτεΐνες ε, για αυξημένη αντοχή σε ζανιοκτώνα που περιέχουν γλυφοσάτη. Για όλου αυτού του λόγου λοιπόν και το σχετισμό της γλυφοσάτη και με, ε, της γλυφοσάτης και ε, να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τη χρήση αυτού του ζυζανιοκτώνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω σημειώσει κάτι εδώ. 16 και στις 20 Μαρτίου του 2016 άκουσα το πιο βάσιμο επιχείρημα και το πιο ζωφερό που ακούστηκε ποτέ σε συνήθειες επιτροπής από τον κύριο Ντες το προσδόκιμο ζωής και πώς θα ζήσουμε περισσότερο δηλαδή για σας το διάρκεια της ζωής δεν είναι πρόβλημα το PCD δεν είναι πρόβλημα γιατί όλοι θα ζήσουμε περισσότερο ο καρκίνος δεν θα μετράει γιατί το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί καμιά νόσος και καμία ασθένεια δεν είναι πρόβλημα γιατί μπορούμε όλοι να ζήσουμε παραπάνω στην εποχή μας να ξεκινήσουμε μια έρευνα για το τι πίνει ο κόσμο στο νερό στην Βαβαρία, γιατί προφανώς κάτι το περίεργο έχει εμφανιστεί σε αυτό το μέρος της Γερμανίας. Εδώ λοιπόν θα ήθελα αυτό πράγματι να καταγραφεί στα πρακτικά Και να συνεχίσω λέγοντας ότι στηρίζω το ψήφισμα αυτό, την αντίρρηση δηλαδή, και ανησυχώ ιδιαίτερως για τις πληροφορίες που έχουμε για τα κατάλοιπα. Νομίζω τα κατάλοιπα στο νερό, το έδαφος, τα τρόφιμα, τα ποτά μας, το ανθρώπινο σώμα, το μετρικό γάλα, ε, είναι προβλήματα σοβαρότατα και πιστεύω ότι ευσταθούν και όλα στα στοιχεία που έχουμε. Δεδομένων των ερωτηματικών λοιπόν που έχουμε, είναι η στιγμή αρχή της προφύλαξης να λειτουργήσει. Και όπως είπαν πολλοί, ε, το γεγονός ότι τα επιστημονικά στοιχεία είναι διαθέσιμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να συμπληρώσουμε τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε ως τώρα γιατί είναι ανεπαρκή και για την μικροβιακή αντοχή ε, στη γλυφοσάτη μεταξύ των ζυζανίων. Βλέπουμε ότι αυτή αυξάνεται διαρκώς, άρα μάλλον έχει τελειώσει η ώρα της της γλυφοσάτης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γιούλικα είναι εδώ και καταλαβαίνω ότι θα έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις για να απαντήσετε. Πράγματι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να απαντήσω. για τα σημεία που έχουν αναπτύξει τα μέλη σας και την ευκαιρία να απαντήσουμε εμείς. Αναγνωρίζουμε και εμείς ότι η γλυφοσάτη αποτελεί ένα, μια πηγή ανησυχίας. Το είδαμε και από τη συζήτηση που έγινε δημοσίω και από τη μελέτη που εκπονήσαμε, διότι εξηγήσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις όλες διαδικασίες. Να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν γέννη βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Τον κανονισμό 1107 του 2009 του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να σεβαστεί. αυτό είναι το πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο εντό του οποίου ε, ενεργούμε και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε με αυτή την ανανέωση ε, και τι έχουμε ένα σκοπό να κάνουμε με τις ε, διαδικασίες ανανέωσης, παράτασης δηλαδή χρήσης αυτής της ουσίας. Στα πλαίσια τη νομοθεσία θεωρούμε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νομοθετικέ διαδικασίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εύρωστε, διαφανεί και σωστέ. Και εδώ επίση ε, εντοπίζονται και το ποιοι πρέπει να πάρουν μέρο στην όλη διαδικασία. Σε αυτή τη φάση να θυμίσω το, την νομοθετική διαδικασία στα τέσσερα βασικά βήματα που προβλέπονται σε τέτοιου είδου περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα θα καταλάβετε και ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς σε καθένα από αυτά τα στάδια. Κατά πρώτον, έχουμε την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών από τα υπεύθυνο κράτος μέλος, το κράτο μέλος εισήγησης, που σε αυτή την περίπτωση είναι η Γερμανία, με τη δική της αρχή προστασίας των τροφίμων. Μετά έχουμε μία ε, αποτίμηση ομοτήμων από την ΕΦΣΑ και όλα τα κράτη-μέλη η οποία εν τέλει οδηγεί στην έγκριση γνωμοδότησης που εγκρίνει η ΕΦΣΑ και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να αναφέρομαι ότι αυτή η διαδικασία εκτίμη αξιολόγηση από τους ομοτήμους οδηγεί σε συμφωνία συμφωνία ε, η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση ε, αφορούσε 27 από τα 27 μέλη, δηλαδή συμφώνησαν ε, οι αρχές των 27 κατών μελών. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης ομοτήμων βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές αλλά και στη βιβλιογραφία, την επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων των συμπερασμάτων της διαδικασίας δημόσιων διαβουλεύσεων μετά την αποτίμηση ε, των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών. Πρόκειται λοιπόν για μια διεξοδική και πλήρη διαδικασία. Ε, μετά από το στάδιο αυτό εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον ε, καταλήγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ και έτσι η αξιολόγηση κινδύνου αποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ετοιμάζεται ένα σχέδιο απόφασης για την παράταση της χρήσης ή την έγκριση μιας ουσίας. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να ανανεώσει την εγκριση μιας ουσιας εδω λοιπον η ευρωπαικη επιτροπη καταληξε στο συμπερασμα οτι μπορει να ανανεωσει την χρηση της ουσίας αυτής. Ε, συζήτησε με τους εμπειρογνώμενες των, των κρατών μελών που ψήφισαν γι' αυτό, απλώς για να το διευκρινίσω, δεν υπήρξε καμία ψηφοφορία ακόμα, διότι είμαστε στην φάση τη διαδικασία λήψη απόφαση. Έχει συζητηθεί λοιπόν η πρόταση με του υπευθύνου των κρατών μελών και να περιορισμεί των συστάσεων χρήση στα κατημέρια. μελη το τέταρτο βήμα είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν επιπλέον ρόλο να παίξουν. Όπως επίσης να επανεκτιμήσουν την εξουσιοδοτήση των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν μπορούν να διευκρινίσουν τις προποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος, προποθέσεις οι οποίες συζητήθηκαν σήμερα εδώ και τις οποίες θα πρέπει να σεβαστούν τα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν ε, απόφαση στοιχεία για τις βοηθητικές ουσίες και για το συνδυασμό των βοηθητικών ουσιών και εδώ είναι ένα βήμα για το οποίο την πλήρη ευθύνη έχουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία εν τέλει θα εξουσιοδοθούν. Όπως προανέφερα λοιπόν, οι βασικοί φορείς εδώ, όπως αναφέρει και η νομοθεσία, είναι τα κράτη-μέλη, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία καθορίζεται έτσι από την νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά την ανανέωση και την παράταση χρήσης της γλυφοσάτης, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2012. Και το Νοέμβριο του 2015 η ΕΦΣΑ κατέληξε στο συμπέρασμα σε κάποια πορίσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν. Αυτό αποδεικνύει κατά την άποψή μου ότι η διαδικασία ήταν πλήρη. Σε αυτό το πλαίσιο ήθελα να θίξω κάποια από τα σημεία, τα περισσότερα σημεία που ακούστηκαν ε, να αναπτύσσονται τα επιχείρηματα των βουλευτών. Θα ξεκινήσω από την αμφιλεγόμενη αξιολόγηση της IARC, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2015. Κατάλαβα ότι στη συζήτηση πήραν μέρο η ΆΕΚ, η ΕΦΣΑ και ο εκτελεστικό διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Επιτροπή σα. Όταν δημοσιεύτηκε η εξολόγηση της ΆΙΑΡΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσως επέκτηνε την εντολή της ΕΦΣΑ από τον Μάρτιο του 2015 κιόλας για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία ελέγχου που έκανε και η ΕΦΣΑ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες για την ταξονόμηση και την κατηγοριοποίηση από την ΆΙΑΡΚ και ότι θα συμπεριλάβει στα συμπεράσματά της την αξιολόγηση αυτή. Κάνοντας κάτι τέτοιο, η ΕΦΣΑ κατέληξε σε άλλο συμπέρασμα από τη ΆΙΑΡΚ. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να εμπιστευτεί πλήρως το στεγανό της διαδικασίας της ΕΦΣΑ, των επιστημονικών πορισμάτων, αλλά και συνολικότερα την όλη διαδικασία με την ε, ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών και την αρχή μιας ανοιχτής διαδικασίας μελέτης ομοτήμων. Να πληροφορήσω την Επιτροπή σας και τα μέλη της, με συγχωρείτε για το βήχα, ότι μετά και από μία άλλη ευρωπαϊκή διαδικασία με θέμα την ταξινόμηση της γλυφοσάτης ανέλαβε δράση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, των Χημικών Ουσιών για, την, ε, για τον έλεγχο και τη μελέτη της κατηγοριοποίησης της γλυφοσάτης ε, σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτή η μελέτη θα περάσει και από μια δεύτερη φάση όπου η γλυφοσάτη θα δούμε αν θα θεωρηθεί καρκινογενής. Η διαδικασία του ΕΚΑΣ επίσης σκοπεύουμε να είναι διεξοδική αλλά μπορεί να είναι και χρονοβόρα και αναμένουμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα σε κάποια φάση στα τέλη του 2017 ή στις αρχές του 2018. Πάντως, εν ώψη αυτής της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη, έχουμε αναλάβει τη σαφή δέσμευση να ε, εγκρίνουμε το πρόγραμμα εξουσιοδότησης κάποιων προϊόντων εφόσον υπάρξει αλλαγή κατηγορίας σε σχέση με την έγκριση ενός προϊόντος. Εδώ να ε, τονίσω ότι σε σχέση με τα στοιχεία που έχει λάβει ο ΕΚΑ και βάσει των πληροφοριών που σήμερα έχουμε, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τον, ε, για τον καρκινογενή χαρακτήρα της γλυφοσάτης σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ε, σε ό,τι αφορά τις τόσο συζητημένες βοηθητικές ουσίες θα ήθελα να ε, θυμίσω ότι εδώ έχουν αρμοδιότητα τα περισσότερα κάτι μέλη και ήδη έχουν αναλάβει δράση για τα μερισμη παραδεκτές χημικές ουσίες. Κάποια κάτι μέλη έχουν κρατήσει κατάλογο με αυτές τις βοηθητικές ουσίες που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τώρα, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπό το φως των ε, ανησυχιών που ακούστηκαν από την ΕΦΣΑ για μία βοηθητική ουσία, την τελοαμίνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ε, σχεδιαστεί σχέδιο κανονισμού, να προταθεί σχέδιο κανονισμού για την απαγόρευση της τάλο αμήνης. Ε, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε, από κοινού με τους εμπειρογνώμες των μελών και της ΕΦΣΑ για να ορίσει κριτήρια και να οριστούν σαφέστερα οι μη αποδεκτοί, οι μη παραδεκτές βοηθητικές ουσίες. Υπάρχει λοιπόν μια μόνιμη επιτροπή που θα μελετά το θέμα των κριτηρίων αυτών και ελπίζουμε να δώσει τα αποτελέσματά της το τελευταίο τριμήνο του 2016. Συγκεκριμένα για τις βοηθητικές ουσίες και ιδιαίτερως για το γλυφοσάτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει επιστήσει την προσοχή των επευθύνων στο θέμα της τάλογαμίνης ε, και το θέμα θα εξεταστεί αναλόγως. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια, ένα επιχείρημα που προβλήθηκε ξανά και ξανά σε αυτή τη συζήτηση, Ε, η διαδικασία ε, εξέτασης ομοτήμων ήδη θεωρείται ομότιμη, μάλλον ομο, ε, διαφανής και ο κανονισμός ορίζει με σαφήνεια ποιες πτυχές και ποια τμήματα των επιστημονικών μελετών πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό. Να θυμόμαστε ότι και η ΕΦΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύονται από την νομοθεσία που οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο ισορροπία από του συνομοθέτε το 2009. Τότε συμφώνησαν οι συνομοθέτε για το θέμα αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κάποιε πληροφορίε όντω πρέπει να δημοσιοποιούνται και έχουν δημοσιοποιηθεί, άλλε θεωρούνται πιστευτικέ και απόρριτε. Ω προς στην περίληψη της νομοδοτησίας μας που δημοσιεύτηκε υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ανεξάρτητη μελέτη όπως έδειξε και η στάση της ΕΦΣΑ σε μια ανεξάρτητη εκδήλωση που χορηγώθηκε από Ευρωβουλευτή από τον κύριο Πότς. Και εμείς θέλαμε να έχουμε πρόσβαση και να αποτιμήσουμε τα επιστημονικά στοιχεία ευρύτερα και όπως ξέρετε ο Επίτροπος Ανδριουκάητης ενημερώθηκε ε, και ε, ανέλαβε δέσμευση να καλέσει τον ανάλογο εμπορικό κλάδο να εκπονήσουν μελέτες ανεξαρτήτως υπό το φως αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης για αυτή τη συγκεκριμένη χημική ουσία. Κάποιοι βουλευτές ε, αμφισβήτησαν, αμφισβήτησαν εμάς και έθεσαν το θέμα των καταλήπων γλυφωσάτης. Να διευκρινίσω ότι ο έλεγχος για τα κατάλοιπα δεν είναι στην, ε, στο πεδίο αρμοδιοτήτων του γραφείου των ε, ζωονόσων και της υγείας των φυτών, αλλά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Βάσει λοιπόν των προγραμμάτων παρακολούθησης των καταλήπων φυτοφαρμάκων, τα πορίσματα δημοσιοποιούνται και με τη συνδρομή της ΕΦΣΑ. Ως προς την γλυφοσάτη, ένα συνολικό πρόγραμμα παρακολούθησης ήδη εφαρμόζεται για τη διάσταση των καταλήπων και ως τώρα έχουμε τουλάχιστον 10.000 δείγματα τροφίμων και ε, διατροφικών προϊόντων με ε, περιεκτικότητα σε γλυφοσάτη που έχουν ε, καθησυχαστικά αποτελέσματα. Από αυτά τα δείγματα το 93% και πάνω δεν έχουν ανοιχνεύσιμα κατάλοιπα καθόλου και μόνον 6,3% αυτών των δειγμάτων έχουν δείξει ανοιχνεύσιμα κατάλοιπα, αλλά και πάλι εντός των νομικών ε, ορίων που έχουν καθοριστεί από το εργαλείο των MRL. Και επίσης μόνο 0,7% έχουν ε, κατάλοιπα πάνω από το επιτρεπτό όριο. Εδώ πρέπει να είμαστε ε, ξεκάθαροι. Δεν σημαίνει αυτή η υπέρβαση των ορίων ε, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Είναι αυστηρός απαραίτητος ε, καθορισμός ορίων για την προστασία των καταναλωτών. Όμως αυτό το ε, ποσοστό από τα δείγματα δεν αποτελούσε ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών. Επίσης για την ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των ε, ζυζανιοκτώνων και την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων τέθηκαν ερωτήσεις. Εδώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό και επενδύουμε χρόνο, πόρους και χρήμα μέσω των προγραμμάτων πλαισίων ε, στην σχετική έρευνα. Συνοψίζοντας, οι επενδύσεις στη σχετική έρευνα και καινοτομία στον τομέα της προστασίας των φυτών, της υγείας των φυτών και της διαχείρισης διαχείριση της ολοκληρωναζής ανιοκτώνων έχει κοστίσει 100 εκατομμύρια στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, στο κεφάλαιο της έρευνας και συνεχίζει να στηρίζεται αυτή η διάσταση και από το Horizon 2020. Έχει λοιπόν γίνει ήδη σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση με πολύ σημαντικούς πόρους που έχουν επενδυθεί σε αυτούς τους ερευνητικούς σκοπούς. Τώρα, ε, γενικότερα, για την αίτηση να υποβληθεί ένα νέο σχέδιο απόφασης. Όπως προείπα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει ένα σχέδιο, μια πρόταση στην μόνιμη Επιτροπή, συζητήθηκε αλλά δεν υπήρξε ψηφοφορία και η συζήτηση θα συνεχιστεί βάσει της τωρινής πρότασης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν τις θέσεις τους και ταυτόχρονα να μας ε, αποστείλουν οποιασδήποτε αλλαγέ θεωρούν απαραίτητες ώστε να ε, στηρίξουν την παράταση της χρήσης ή όχι της γλυφοσάτης. Η Ευρωπαϊκή λιποσατης η επίσης κατέστησε σαφές ότι ε, θέλουμε την συνολική στήριξη των κρατών για το θέμα αυτό και πραγματικά το σχέδιο κανονισμού θα συζητηθεί σε μία από τις επόμενες, τις επερχόμενες συναντήσεις της μόνιμης επιτροπής. Έγινε πολλή λόγος και για την αρχή της προφύλαξης σήμερα. Όπως προείπα και όπως προτώνησα, Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματικά πλήρη εμπιστοσύνη στου φορεί που εμπλέκονται σε αυτή την επίσημα καθορισμένη διαδικασία, τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν τι αρμόδιε αρχέ του, του φορεί αξιολόγηση κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και στην ΕΦΣΑ. Όπω είπα, η διαδικασία είναι ευρύτατη. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αξιολόγηση κινδύνου για την γλυφοσάτη και η ενδυνάμει ανανέωση και παράταση χρήσης της, ε, παράταση της χρήσης της ήταν βασιμότατη και δεν υπάρχουν λόγοι διαχείρισης κινδύνων που να επιβάλλουν κάτι διαφορετικό. Για να είμαστε σαφείς στην πρότασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει αυτό το πλαίσιο, τη σχετική απόφαση, εφόσον η διαδικασία ή τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Ουσιών που εξετάζουν το καρκινογόνο της γλυκοσάτης δείξουν ότι υπάρχουν αποδείξεις ή ενδείξεις για κίνδυνο στη δημόσια υγεία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση θα ξαναδεί την ε, αδειοδότηση, την παράταση χρήση τη γλυφωσάτη. Αλλά άμα δεν υπάρξουν σαφεί ενδείξει. Ε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αναλόγως όμως με τα τι στοιχεία μπορεί να προκύψουν, ανά πάσα στιγμή μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ενεργοποιήσει τη διαδικασία της ε, αναθεώρησης, της επανεξέτασης της παράτασης ε, χρήσης. Νομίζω, άσχετα με την περίοδο που κρατάει αυτή η παράταση, 15 χρόνια, νομίζω ότι θα απάντησα τα περισσότερα, απλώς κλείνοντας να αναφερθώ στο θέμα της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κατ' επέκταση στην όλη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει για τη σημασία της εμπιστοσύνης ε, προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ακολουθώντας το συμπεφωνημένο νομοθετικό πλαίσιο κάνουμε ένα πολύ σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ακριβώς έτσι δημιουργούμε και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Ακολουθώντας λοιπόν έτσι την ιωθώσα διαδικασία όπως προβλέπετε εμπλέκοντας όλους τους υπευθύνους και επιστημονικούς φορείς που ε, ε, είναι αρμόδιοι βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, φροντίζουμε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη την εκπόνηση ανεξάρτητων μελετών από την ΕΦΣΑ, αλλά και τη δυνατότητα των κρατών μελών και των αρχών τους να κάνουν τα δέοντα. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός λόγος να διατηρηθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης και όπως προείπα η εμπιστοσύνη στην ΕΦΣΑ είναι ακρογωνιαίο λήθος στο όλο σύστημα. Με αυτά θα ήθελα να πάψω, ε, να ολοκληρώσω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρόνο, γι' αυτό δεν θα σχολιάσω όλο όσο μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα αντιδράσω αυτά που είπε ο κύριος Δες, γιατί είναι αδύνατο να μην αντιδράσει κανείς. Αυτή η πρόταση ε, για την αντίρρηση δεν ε, εκπορεύθηκε από καμία μη κυβερνητική οργάνωση εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά από μένα και από συναδέλφους. Λυπούμε που δεν ήσταν παρόν στην επιστημονική διάσκεψη. Αλλά πραγματικά ήταν ένα από τα μόνα αυτά που άκουσα, και αυτό δεν μπορούσα παρά να σχολιάσω. Παίρνουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη την εξέταση του σχεδίου έκθεση γνωμοδότηση ε, τη Επιτροπή Περιβάλλοντο σχετικά με την εφαρμογή τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε, ιδίω όσον αφορά τι καταληκτικέ παρατηρήσει τη Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, CRPD. Η συγγετριά μας είναι η κυρία Νέσα Τσάιλτερς που συνέταξε για την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων γιατί ε, πολλές ε, επιτροπές συνεργάστηκαν για τη σύνταξη της γνωμοδότησης και βοηθώ ε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους και τους βοηθούς αλλά και τη γραμματεία γιατί είχαμε πολύ στερές προθεσμίες. Με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με, αναπηρία το 2010 ήταν ε, ένα ορόσημο γιατί ήταν η πρώτη διεθνής συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλους τους συμπολίτε μας η αξιοπρέπεια είναι εγγενές θέμα και η αναγνώριση διασφάλιση συμμετοχή και πλήρη ένταξη στην κοινωνία απαραίτητη και κατοχυρώνεται στο πρωτογενέ ευρωπαϊκό δίκαιο και σε πολλά νομοθετικά εργαλεία όπω είναι η ελόγω σύμβαση του ΟΗΕ. Στην πράξη βέβαια, άνθρωποι με αναπηρίε. Μια στιγμή, παρακαλώ, λίγη ησυχία αγαπητοί συνάδελφοι. Όσοι θέλουν ε, να, μιλήσουν, ας εξέλθουν από την αίθουσα γιατί έχουμε δουλειά. Στην πράξη όμως άνθρωποι με αναπηρίες 80 ε, περίπου εκατομμύρια συμπολίτε μα αντιμετωπίζουν δυσκολίε και φραγμού και δεν μπορούν να απολαύσουν πλήρω τα δικαιώματά του. Όπω προβλέπετε για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τη σύμβαση, μια αρχική έκθεση εφαρμογή έγινε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2014 με ε, επίσημη ανταλλαγή απόψεων ε, στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν οι καταληκτικές παρατηρήσεις τη Επιτροπής του ΟΗΕ ε, επί της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, και μάλιστα η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει μετά το καλοκαίρι. Ε, πριν από την επίσημη αυτή απάντηση. Η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Θεμάτων ετοιμάζει την σχετική έκθεση, εξού και η δική μα γνωμοδότηση για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση τη έκθεση αυτή. Γιατί μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα τη πρόσβαση σε ποιοτική ε, υγειονομική και ιατρική περίθαλψη για του ανθρώπου με αναπηρίε. Οι αναπηρίε δυστυχώ σχετίζονται στενά με κακή υγεία και δυσχέρειες και εμπόδια προσβασιμότητας. Μπορεί για μερικούς να είναι θέμα κληρονομικό η κακή υγεία, αλλά τουλάχιστον δεν θα πρέπει να επιδεινώνεται από ελλειπή πρόσβαση σε ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, που δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά σε μια καταξινόμηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για τις δυσκολίες ε, και τους διάφορους τρόπους διακρίσεων, στους οποίους υπόκεινται πιο ευάλωτοι συμπολίτε μας που έχουν αναπηρίε ε, και ήδη αρκετέ δυσκολίε στη ζωή του εξαιτία του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται η κοινωνία σε αυτούς. Οι γυναίκες με αναπηρίε, για παράδειγμα, έχουν υψηλότερα ποσοστά κακής υγεία και ο γυναικείος πληθυσμός έχει και προβλήματα ψυχικής υγεία ε, πάνω από το μέσο όρο και μάλιστα ιδιαίτερα στις μετανάστριες ε, είναι πολύ πιο ψηλά αυτά τα ποσοστά. Θα πρέπει να δούμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της αναγνώρισης της ισότητας των δικαιωμάτων στη θεωρία και τις σημαντικές διαφορές ε, που υπάρχουν στην πράξη λόγω κακής ε, μεταχείρισης ή ανεπαρκούς προσφοράς ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης οι διαφορές στο επίπεδο ποιότητας ε, της ιατρικής περίθαλψης ε, για τους, ε, για τους αναπήρους σε σχέση με τους μη ανάπηρους προϋποθέτει σωστή κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Γιατί η προσέγγιση που έχουμε στην φροντίδα των ατόμων με αναπηρία θα εξαρτηθεί και από διάφορες ε, κοινωνικές οργανώσεις και οι παραδοσιακές νομικές ε, ε, απόψεις για την δικαιοπρακτική ικανότητα μερικές φορές άδικα στερούν από κάποιους ανθρώπους το δικαίωμα υπολογής γιατί η ενημερωμένη συνένεση είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε ίση ε, πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική και περίθαλψη. Και φυσικά αναπηρία δεν σημαίνει ε, ακούσια, ακούσιο αγγλισμό και κακή μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή μητροπή να μεριμνήσει για τα άτομα αυτά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την σωστή ε, και ποιοτική πρόσβαση. Ε, οι γυναίκες ε, ε, υπόκειται σε πολύ μεγαλύτερη παραβίαση των δικαιωμάτων τους όπως αναγνωρίζονται στις ευαίσθησες Βιέννης. Και η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι σημαντικός κίνδυνος. Επίσης η στήρωση ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική επέμβαση θα πρέπει να υπόκειται στο, στην συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Αυτά θα πρέπει να καλύπτουν και τον οικογενειακό σχεδιασμό και την αναπαραγωγική υγεία. Δεν θα πρέπει να υστερήσουμε σε σχέση με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία, η νομοθεσία μας. Και αυτό προϋποθέτει και την διασυνορική παροχή ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης. Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, διορθώσουμε τα κενά με πανευρωπαϊκές κατευθυντήρε γραμμές και προσιτέ πληροφορίε σε όλους, ακόμη και στους ανθρώπου, με αναπηρίε, που χρειάζονται ενημέρωση σε συγκεκριμένες μορφές γιατί δεν θα πρέπει ένας, ένα άτομο με αναπηρίες να υποστεί περαιτέρω διακρίσεις. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να μας υποχρεώσει να αναλάβουμε και το κόστος για να εκπληρώσουμε τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, καλύτερη πρόσβαση σε ε, ηλεκτρονικές, ε, ηλεκτρονική για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλους. Αυτά όλα θα πρέπει να τα κοιτάξουμε ώστε να αποφύγουμε και διατομιακή διάκριση. Σε ό,τι αφορά τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρίε, γυναίκε, παιδιά, ΛΟΑΔΜΑ ή μετανάστε, ε, είναι πιο ευάλωτε ομάδε. Αλλά είμαστε μέλη μια κοινωνία που θα πρέπει να περιθάλπει και να βοηθά όλα τα μέλη τη. Γι' αυτό και θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους τα δικαιώματα που καθορίζουν τον πολιτισμό, τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Εκ μέρους του ΕΛΚ, το λόγο και ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Τσάλντες για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Το σχέδιο κειμένου είναι πολύ ισορροπημένο, καλύπτει όλα τα βασικά ζητήματα και αποτελεί πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Σύντομα θα προσπαθήσω να αναφέρω τα θέματα που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε αυτό που δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες ε, συστηματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, στην πρόσβαση ε, στην υγεία από ό,τι άλλη. Αυτή η ανισότητα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον, στην αυτόνομη διαβίωση των ανθρώπων αυτών ε, και σε ίση βάση με άλλους. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε ε, εξίσου καλή πρόσβαση στην υγεία συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με πιο συντονισμένο τρόπο και να συμπληρώνονται από εθνικά μέτρα όπου είναι απαραίτητο ως μέσο βελτίωσης ε, του ε, επίπεδου διαβίωσης των ανθρώπων με αναπηρίες. Για τα μέτρα αυτά η ευθύνη εναπόκειται στα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την προσβασιμότητα στα συστήματα υγείας για τα άτομα με αναπηρία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη όσον αφορά τον, ε, την ε, συγκέντρωση των δικτών για τον χρόνο αναμονής και άλλες στοιχείες που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των ανθρώπων με αναπηρίες. Επίσης, όσον αφορά την ε, εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, θα πρέπει να εξετάζεται και η δυνατότητα των ανθρώπων με αναπηρία να εποφελούνται από την οδηγία αυτή με τον ίδιο τρόπο με ανθρώπους χωρίς αναπηρίες. Για τα άτομα με αναπηρία μπορεί να ε, να απαιτούνται επιπλέον δαπάνες ε, και τα κράτη-μέλη να μην είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν τις δαπάνες αυτές στον ασθενή. Επίσης, θα πρέπει να εκπονηθεί η έκθεση προόδου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τζούλη, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε σε αυτά που είπε το Ελκ και η συγκήτρια. Θέλουμε να την, ευχαριστούμε για, να την ευχαριστήσουμε για την έκθεσή της που πιστεύουμε ότι καλύπτει όλα τα θέματα που θα πρέπει να καλύψουμε. Ε, προσθήκη θα κάνουμε μόνο σε ένα σημείο που έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Στην έκθεση υπάρχει η αρχή της προσβασιμότητας. και της ε, πλήρη επιγνώσης συγκατάθεσης, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να αναπτύξουμε τις διαδικασίες ώστε αυτό να είναι εφαρμόσιμο στην πράξη, όπως ε, είναι και το θέμα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Θα πρέπει να προσέξουμε να φροντίσουμε να υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ εξαιρετικά. Χωσέ Ινάσιο Φαρία από το Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά τη για την σύνταξη αυτού του σχεδίου νομοθεσής, για την περίπτωση αυτών των ανθρώπων με αναπηρίες Πρέπει να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, με αναπηρίε. Όμω πρέπει να εντοπίσουμε και του τομεί που πρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματά του ανεμπόδιστα τα άτομα αυτά και τομεί που χρήζουν ιδιαίτερη προστασία. Η κύρωση τη σύμβαση αυτή από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρηθεί οπωσδήποτε ω μια θετική κίνηση. Και έχει εντείνει την ε, ε, δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα άρθρα 21 και 26 τη Χάρτα των Απελευθερών Δικαιωμάτων για την προστασία των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίες, εξασφαλίζοντα τη συμμετοχή τους με τρόπο ισότιμο και πλήρη σε όλε τι δραστηριότητε τη κοινωνία. Θέλω λοιπόν να στηρίξω και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ε, την, ε, την εισηγήτρια που είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό, για την έκθεση που υπέβαλε. Και την περίοδο προγραμματισμού του 2014-2020 και για την χρηματοδότηση που προβλέπεται από τα διευθυντικά ταμεία και τα ταμεία ανάπτυξης πρέπει να ε, προάγουμε την ε, μη διακριτική μεταχείριση και την συμπεριλήψη σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας των ανθρώπων της, ε, με ειδικές ανάγκες για να ικανοποιήσουμε και τους στόχους της σύμβασης. Πρέπει λοιπόν να επιχειρήσουμε ακριβώς τέτοιες σχετικές δράσεις και η γνωμοδότηση σωστά θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία μνήα για την εκπόνηση συγκεκριμένων πολιτικών για τα παιδιά και τους εφήβους που έχουν ε, ε, συγκεκριμένες ειδικέ ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη το τι χρειάζονται αυτά τα παιδιά και εφηβοί και πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το δρόμο τους προς την σωστή ανατροφή, ανάπτυξη και αγωγή προς όφελος της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας. Πρέπει να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση και την γνώση του πληθυσμού για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και την ε, προστασία των παιδιών αυτών και των εφήβων, για την νοητική, ψυχολογική και ε, πνευματική τους υγεία και για την πλήρη του συμπερίληψη. Ε, επίσης μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρταση κατάρτιση και στηρίξη των ανθρώπων που μπορεί να έχουν ειδικέ ανάγκες. Το αριθμός κλήσης 72 112 δεν είναι ε, ο αριθμός λοιπόν 112 και όλες οι πολιτικές ε, που θα σχεδιάζονται θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη το τι ιδιαίτερα χρειάζεται να προβλεφθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμη και όταν πρόκειται για περιοχές αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων. Ε, πρέπει να αναλυθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και πάντοτε με την ε, συγκατάθεση των ατόμων αυτών. Το ίδιο και για την ποιότητα των πρώτων υγεία που προφέρονται στα, στα άτομα αυτά. Θα πρέπει σε όλε τι φάσει να σχεδιάζονται υπηρεσίε και προϊόντα στον τομέα τη υγεία για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε που να είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στι δικέ του ε, ανάγκε για να διασφαλίζουμε την προστασία και την ασφαλεία του. Πρέπει να σκεφτούμε την ε, προσέγγιση κόστος ωφελία, την ε, στιγμή οικονομική εξέταση των προϊόντων αυτών στην ε, κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων αυτών. Αναπομονώ για τη συνεργασία με τους συναδέλφους στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, μάλλον είναι η πρώτη φορά που ε, μας περιμένουν εμά οι συντονιστές και όχι εμείς τους συντονιστές. Συνεχίζω λοιπόν στα τσεχικά για να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Κατερίνα Κονέτσνα. Ευχαριστώ. Ο χρόνος περνάει, γι' αυτό θα είμαι λακωνική, μια και οι συνάδελφοι με κάλυψαν σε πολλά σημεία. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη συντάκτρια της γνωμοδότησης ε, για την πρότασή της, που είναι πολύ κοινωνικά ευαίσθητη. Και θεωρώ ότι οι τροπολογίες μας ε, θα επισημάνουν περαιτέρω τις κοινωνικές πτυχές αυτού του ζητήματος. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην παράγραφο 4 θεωρώ ότι ως Επιτροπή θα πρέπει να τονίσουμε τη σχέση που έχει η, προσβασιμότητα, η ποιότητα, οι προσιτές τιμές και η διαθεσιμότητα. Θα πρέπει η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα να λαμβάνουν υπόψη τις τιμές που μερικές φορές είναι πολύ ψηλές. Θα πρέπει να είναι δωρεάν η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για τους ατόμους με αναπηρίες. Θα πρέπει επίσης ε, η φροντίδα της υγείας να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και να μην τους επιβαρύνει περαιτέρω. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Περιμένω τις τροπολογίες για να τις εξετάσουμε. Πάντως σίγουρα το σχέδιο είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Ντορνανό από την ομάδα των Εθνών και των Ελευθεριών. πολλέ παρατηρήσει για την γνωμοδότηση. Καταρχήν έχουμε τη διαπίστωση ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ αναπηρία και κακή υγεία. Νομίζω ότι αυτή είναι ταυτολογία πλεονασμός ε, που προκύπτει από τον κανονιστικό πληθωρισμό των κειμένων. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, είμαστε πιο συνοπτικοί και άρα και πιο ευανάγνωστοι. Και παρόλο που οι άνθρωποι με αναπηρίε έχουν προβλήματα πρόσβαση, αυτό είναι αλήθεια, το να μιλήσουμε για φραγμό στι υπηρεσίε υγεία, αυτό είναι υπερβολικό. Γιατί κάτι τέτοιο προποθέτει μια σκεμμένη δράση. Επίση, τα ψυχικά προβλήματα, ε, θέματα γενετήσια ταυτότητα και η μετανάστευση και η συμπερίληψη και των τριών σε ένα τέτοιο θέμα νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Επίσης, ε, ε, το θέμα της ε, λογικής μεταρρυθμίσης για ή μάλλον διαρρύθμισης. δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε μεγάλο κόστος επιχειρήσεις για τέτοιους είδους διαρρυθμίσεις για να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να δίνουν πληροφορίες σε όλους και στους ανθρώπους με αναπηρίες και νομίζω ότι είναι υπερβολικό να ε, περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει το δυναμικό της τηλεϊατρικής ε, και να ε, εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευέ στους ανθρώπους με αναπηρία. Θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στις καινοτομίες, αλλά δεν θα υποκατασταθεί σε αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Ή δεν έχουμε εκπρόσωπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα δύο πράγματα να κάνω στην παρέμβασή μου. Καταρχάς να επαναλάβω την αφοσίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των συμπερασμάτων της ε, του Οργανισμού της, Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το σχέδιο γνωμοδότησης και που θίγει το θέμα της σημασίας της ίσης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα και με την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια δεν θέλει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Δεν θα προσθέσω πολλά. Όλα όσα ακούστηκαν ήταν πολύ χρήσιμα και δεν μας μένει πολύ χρόνος. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα ήθελα να πω στην κυρία Ντορνάνο ότι φάνηκε να μιλάμε ως αν τα εμπόδια στην προσβασιμότητα να ε, έχουν τοποθετηθεί εσκεμένα. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται για συνωμοσία, αλλά είναι κάτι που γίνεται στην πράξη και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 23 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ 26 Απριλίου, στην Επιτροπή ΕΜΠΛ 30 Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο του 2016 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στις 9 για τις ψηφοφορίες.